συνεχίζουμε την απογευματινή συνεδρία μας, η οποία αρχίζει με ακρόαση για τις ξένες άμεσες επενδύσεις, μεταβατικές ρυθμίσεις και μελλοντική ευρωπαϊκή διεθνής επενδυτική πολιτική. Η συνθήκη της Λισαβόνας ε, πηρέασε την... Ε, ε, τις εξελίξεις και τις αρμοδιότητες της Ένωσης και μπορεί να γίνει πολύ σημαντικό μέσον που θα διέπει τις εξωτερικές σχέσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γίνεται τώρα συνομοθέτης και ε, θα πρέπει να εκδίδει σύμφωνη γνώμη πριν από οποιαδήποτε επενδυτική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών. Η Επιτροπή μας έχει, είναι υπεύθυνη ε, να εξετάσει δύο εκθέσεις για το επενδυτικό πακέτο της Κομισιόν. Έχουμε την έκθεση Καρλ Σλούτερ για την πρόταση σχετικά με τις μεταβατικές ρυθμίσεις για τα BIT, τα BITS, είναι εδώ ο κανονισμός για την πατρογονική ρήτρα, όπως λέμε, grandfathering, και μια άλλη για το μέλλον της ε, επενδυτική πολιτικής της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε σχέση με αυτές τις δύο εκθέσεις υπάρχουν πολλές προκλήσεις και για μας, από πολιτικής και νομικής άποψης. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να διοργανώσουμε μια ακρόαση και έχω την χαρά να σας παρουσιάσω τους ομιλητές μας που είναι όλοι διακεκριμένοι. Πρώτα έχουμε τον δόκτωρα Στέφαν Γουλκοκ, λέκτορα στο London School of Economics. Ήμουν και εγώ φοιτητής εκεί στη δεκαετία του 70 Ο δόκτωρ Γούλκοκ επίσης ε, ήταν ε, επικεφαλής του έργου για τις ε, άμεσες ξένες επενδύσεις. Δεύτερον, η κυρία Ναταλή Μπερνασκόνη Όστερ Βάλτερ, η οποία είναι νομικός και επικεφαλής του προγράμματος του, των επενδύσεων από του Διεθνούς Ινστιτούτου Αϊφόρου Ανάπτυξης στη Γενέβη, Ελβετία, ο δόκτωρ Κρίστιαν Τίτιε, ο οποίος είναι καθηγητής Δημοσίου Ευρωπαϊκού Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Διευθυντής του Ινστιτούτου Οικονομικού Δικαίου στην έδρα, στη σχολή, ε, στη νομική ε, ε, σχολή, στη σχολή Οικονομίας και Επιχειρήσεων στο Μάρτιν Λούθερ Πανεπιστήμιο στο Χάλε Βίτεμπεργκ στη Γερμανία και ο, δο, ο κύριος Άντριαν Βάντερ Χόφεν, ο οποίος είναι Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων στο Business Europe. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ πλούσιο το βιογραφικό των ομιλητών. Ο, κύριος Μάουρο Πετριτσόν εκπροσωπεί την ε, Κομισιόν, είναι ε, διευθυντής ε, ε, στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Θα δώσω με το λόγο στους προσκεκλημένους μας. Παρακαλώ όλοι να τηρήσουν το, τα 10 λεπτά. Θα υπάρχει δυνατότητα να δευτερολογήσετε κατά την διάρκεια των έρωτα απαντήσεων που προβλέπουμε αργότερα στη συζήτηση. Προχωρούμε λοιπόν με τη σειρά της παρουσίασης και δίνω πρώτα το λόγο στον δόκτωρα Στέφαν Γουλκοκ. Να τον καλωσορίσω και να τον διαβεβαιώσω ότι είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς που έχουμε τη χαρά να τον ακούσουμε. Ευχαριστούμε που ήρθατε, έχετε το λόγο. Ο στόχος μου σήμερα είναι να κάνω μια εισαγωγή για τα θέματα κλειδιά που θα συζητηθούν από την Επιτροπή, την Επιτροπή σας. Η συμπερίληψη των ξένων της πολιτικής εισαγωγών ε, έχει ως χαρακτηριστικό την πρόσβαση των ευρωπαϊκών εταιριών, ή την ενίσχυση της πρόσβασης στην αγορά και την επιρροή τους σε έναν τομέα ο οποίος υφίσταται μετασχηματισμό. Μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είχε ρυθμίσεις και κανόνες άμεσους που επηρέαζαν είτε τα κράτη-μέλη είτε συνθήκες ε, ε, διμερείς με τα κράτη-μέλη είτε διάφορα, διάφο, συμφωνίες άλλου τύπου. Τελικά, στην συνθήκη δεν έχουμε ε, λεπτομεριακή έκθεση ε, των τεκτενομένων και αυτό δίνει πολλές δυνατότητες ερμηνείας για τις άμεσες ξένες επενδύσεις ε, και για τις αποκλειστικές αρμοδιότητες, για τις υποσχέσεις για αποκλειστικές αρμοδιότητες της ΕΕ. Πρέπει λοιπόν ένας τρόπος προσέγγισης ε, στις διαπραγματεύσεις της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις αρμοδιότητες της ΕΕ είναι αυτός που υπήρξε στο παρελθόν η πρόσβαση στο εμπόριο ή υπάρχει σήμερα ε, και η σχέση με τις επενδύσεις. Η Επιτροπή προσπαθεί να βρει εντολές για να συμπεριλάβει στα, τις επενδύσεις και αυτό είναι κάτι το οποίο το εξετάζουν οι επιτροπές ως ε, περιεχόμενο της οποιασδήποτε συμφωνίας επί των επενδύσεων μελλοντικής ε, συμφωνίας. Η πολιτική της ε, ΕΕ αφορά τους εταίρους που αναζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικά, ευρύτερα μπορούμε να πούμε ότι η μελέτη προκύπτει από την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα κριτήρια της ταύτισης και ευθυγραμμίζεται με την πολιτική της ΕΕ με όρους της ε, Καθολικής Ευρώπης και όρους τους οποίους εξέθεσε ο Επίτροπος Δούρκοπτο στην πρωινή συνεδρίαση στο λόγο που εκφώνησε. Έχουμε την, το δυναμικό της αγοράς ως προϋποθέσεις, την προβλεψιμότητα της εφαρμογής των επενδύσεων και ε, υπάρχει ε, μια δυνατότητα για τους ε, διαπραγματεύοντες τα θέματα αυτά να ε, προσαρμοστούν στα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ακόμα και η Ρωσία εστιάζεται σε συμφωνίες ε, γενικές για ξένες επενδύσεις. Αυτό συμπεριλαμβάνει και τον Καναδά, τη Σιγκαπούρη και την Μαλαισία ε, σε ε, συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου. Αυτές είναι και οι συμφωνίες οι οποίες αυτή τη στιγμή γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Ε, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει πανεπιστημιακή φιλολογία σε σχέση με αυτές τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου και επενδύσεων. Υπάρχουν οπωσδήποτε οι κατηγορίες των FTAs, δηλαδή των ε, συμφωνιών ελευθερού ε, εμπορίου. Υπάρχουν οι διμερείς συμφωνίες επενδύσεων, οι οποίες έχουν μια σάφια γενικά και αυτό χαρακτηρίζεται σε όλη τη σχετική φιλολογία. Ένα από τα θέματα κλειδιά είναι ότι η συζήτηση εστιάζεται πολύ συχνά στο επίπεδο της προστασίας των επενδύσεων. Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες, αν απλουστεύσουμε κάπως την συζήτηση. Καταρχήν, ε, οι επιλογές ένα, να υπάρχουν ε, ευρύτερες προδιαγραφές προστασίας, δηλαδή να ακολουθηθεί το μοντέλο των περισσότερων κρατών μελών που προσφέρουν μεγαλύτερη προστασία και έχουν την δυνατότητα να παράσχουν υψηλό επίπεδο προστασίας στους Ευρωπαίους επενδυτές αλλά αφήνουν ένα ευρύ πεδίο για ερμηνεία, για το επίπεδο της προστασίας και αυτό το επίπεδο ερμηνείας το διαχειρίζονται διαιτητικά δικαστήρια. Η δεύτερη επιλογή είναι να υπάρχει ένας πιο συγκεκριμένος ορισμός ε, για να μπορέσει να διευκρινίσει τα επίπεδα των προδιαγραφών της προστασίας και να αφήσει λιγότερο χώρο για ερμηνεία στα δικαστήρια ή σε άλλα αρμόδια σώματα και να αυξήσει τον δημόσιο έλεγχο ε, στον, στο δίκαιο των ε, ξένων επενδύσεων και στη διατησία τους δεν νομίζω ότι έχουμε ώρα για να τα δούμε τα θέματα αυτά λεπτομεριακά, αλλά θα ήθελα να φωτίσω ορισμένα στοιχεία κλειδιά λίγο περισσότερο. Οι περισσότερες ε, συμφωνίες μιλάν για μη διάκριση, δηλαδή η Εθνική ε, Συμφωνία ε, συζητάει για το αν θα υπάρχει πρόσβαση αν θα ελαμβάνεται η απόφαση από την κυβέρνηση ή αν θα υπάρχει καλύτερη πρόσβαση στις αγορές. Ένα πρόβλημα που τέθηκε ε, είναι ότι υπάρχουν ε, ορισμένες απαιτήσει από τα πιο ευνοούμενα κράτη ή ε, παραδείγματος χάρη η εθνική διαχείριση, μεταχείριση Οπότε έχουμε ε, ένα πρόβλημα ερμηνείας για τη μία ή για την άλλη κατηγορία. Ένα άλλο κλειδί θέμα είναι η δίκαια και ισομερής μεταχείριση η οποία βασίζεται σε ορισμένες προδιαγραφές. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν θα γραφεί απλώς ότι θα υπάρχει δίκαιη μεταχείριση, αν θα γραφεί αυτό στη συμφωνία ή αν θα δοθούν πιο συγκεκριμένες προδιαγραφές περιγραφόμενες μία προς μία. Ε, μετά έχουμε το επόμενο θέμα, το επόμενο σημαντικό θέμα, ποιος ορισμός ε, έμεσης απαλωτρίασης είναι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εάν εξετάσετε τα υπάρχοντα κράτη-μέλη βλέπετε ότι τα περισσότερα από αυτά στην ε, μελέτη που κάναμε είδαμε τα τελευταία ε, κράτη-μέλη, τα τελευταία 15 κράτη-μέλη τα πιο πρόσφατα συμπεριέλαβαν τα περισσότερα διάφορα μέτρα για τις απαλωτριώσεις ενώ άλλα από αυτά η Ιταλία ας πούμε και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είχαν τέτοιου είδους ε, προβλέψεις για διμερείς συνθήκες επενδύσεων. The, uh, one controversial issue in investment. Έχουμε λοιπόν ένα άλλο πρόβλημα, ε, το πρόβλημα της διατησίας το οποίο τίθεται ταυτόχρονα και αποτελεί μέρος των θεμάτων κλειδιών, δηλαδή τι προσέγγιση να έχουν τα κράτη-μέλη, με ποια συμφωνία. Μπορεί βεβαίω κανείς να ρωτήσει αν θα πρέπει να υπάρχει καν μια τέτοια συμφωνία και αν δεν θα πρέπει να συμπεριλάβει καθόλου την οποιαδήποτε συμφωνία ε, της ΕΕ για επενδύσεις. Θα είναι τότε πολύ πιο αδύναμη, θα είναι, δεν θα έχει καμία σχέση, θα είναι άσχετη ύστερα ε, έχουμε πιο ουσιαστικές ερωτήσεις, ε, ποιο βαθμό διαφάνειας θα πρέπει να αναζητήσουμε στις ε, εργασίες διατησίας, πώς θα μπορούσαμε να αποφύγουμε τις πολλαπλές προσφυγές και τις εντελώς διαφορετικές ερμηνείες του νόμου και πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε αναθεώρηση ή έφεση για τις αποφάσεις των διαιτητικών δικαιωμάτων δικαστηρίων. Ορισμένες ε, ε, τέτοιου είδους ε, επενδύσεις, αιτήσει για επενδύσεις προβλέπουν και μία ρήτρα η οποία μιλάει για τις διαιτητικές αποφάσεις και για το θέμα της προσφυγής ή της αναθεώρησης. Υπάρχουν ύστερα διμερείς συνθήκες, οι μεταβατικές ρυθμίσεις. Ε, σχετικά με τις ε, ε, πολιτικές της ΕΕ. Στον τομέα αυτό το σημαντικό είναι το πώς θα αντιμετωπιστούν αυτά τα πολύ σύνθετα νομικά θέματα, τα οποία όταν συζητούνται έχουν πολύ διαφορετικές δυνατότητες. Για τον κανονισμό προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να υπάρξει μια γενική παροχή ε, αδειών ε, για τα, στα υπάρχοντα κράτη-μέλη, στα οποία να δίδεται αυτή η δυνατότητα και υπάρχει και η μεταβατική περίοδος, γιατί οι αρμοδιότητες οι οποίες ε, τους δίνονται, δίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έτσι η νομική βεβαιότητα αποδυναμώνεται ε, και υπάρχει η δυνατότητα να αποσυρθεί η άδεια, απόσυρση της άδειας σύμφωνα με το άρθρο 5.1 ε, αυτό είναι, ανήκει στον κανονισμό που λέει ότι η απόσυρση των αδειών στην περίπτωση που μία άδεια δεν ακολουθεί την ουσία της ε, πολιτικής. Δηλαδή αν θέλει να διαπραγματευτεί μια ε, σύμβαση με την Κίνα η ΕΕ για επενδύσεις ε, και στην περίπτωση αυτής της διαπραγμάτευσης υπάρχουν ερωτήματα. Το θέμα είναι πώς θα δοθούν απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα και δίδονται ορισμένες απαντήσεις είτε να απορριφθεί ο κανονισμός γιατί δίνει πάρα πολλές εξουσίες και αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Υπάρχει όμως και η δυνατότητα της ε, έγκρισης του ε, η οποία θα πάρει πάρα πολύ χρόνο στα δικαστήρια. Είναι λοιπόν πάρα πολύ χρονοβόρα και θέτει ένα αμφιβόλο την νομική βεβαιότητα με τη σειρά της. Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα καταθέσεως τροπολογιών η οποία αναγνωρίζει οποιαδήποτε αποδυνάμιση της προτάσεως δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέρη ακόμα και να, μπλοκάρουν την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής στον τομέα αυτό. Χρειάζεται λοιπόν να βρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα στις διαφορετικές αυτές αντιμετωπίσεις. Εναλλακτική λύση είναι να εστιαστούμε στην λήψη αποφάσεων, δηλαδή να βρούμε μια διαδικασία λήψης αποφάσεων η οποία δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα φοραμένα μέρη να έχουν ε, ικανοποίηση, να, να έχουν ικανοποιητικές πολιτικές οι οποίες να συμφωνούν με τα γενικά συμφέροντα της ΕΕ. Ως συμπέρασμα λέμε ότι η εμπειρία στην πολιτική εξωτερικού εμπορίου της ΕΕ ε, προτείνει να υπάρχει μια αποτελεσματική πολιτική η οποία αναβασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και ενδιαφερόντων και αυτό διευκολύνει την οικοδόμηση ενός νομικού πλαισίου και, ε, και δεν χρειάζεται έτσι μια πολύ σύνθετη νομοθεσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε καθηγητά για την παρουσία σας. Σας περάσουμε στη δεύτερη ομιλήτρια, την κυρία Ναταλή Μπερνασκόνη Αστερβάλντερ. Δέκα λεπτά και πάλι έχετε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Στη σύντομη παρουσίασή μου θα επικεντρωθώ στο θέμα της προστασίας των επενδύσεων και από αυτό εννοώ το στοιχείο της μεταγκατάστασης των διεθνών επενδυτικών συμφωνιών θα δούμε καταρχήν ορισμένε από τι ε, τάσει ε, στον τομέα τη προστασία ε, των επενδύσεων και τη διευθέτηση διαφορών και μεταξύ άλλων θα δούμε ότι η Ευρώπη, όπω και άλλα τμήματα του κόσμου, ήδη αντιμετωπίζουν ένα αρκετά μεγάλο αριθμό διευθετήσεων επενδυτικών συνθήκων και στη συνέχεια θα δούμε κάποιε από τι κύριε προκλήσει που έχουν καταστεί εμφανεί στον τομέα τη επενδυτική προστασία ε, και θα εξετάσουμε ζητήματα που έχουν προκύψει σε σχέση με του ουσιαστικού κανό, ουσιαστικού δικαίου που συμπεριλαμβάνονται στι επενδυτικέ συνθήκε, ε, όπω και στο μηχανισμό επίλυση διαφορών και θα αντλήσουμε εμπειρίε και από άλλε χώρε όπω είπα και ο Καναδά και θα εντοπίσουμε τρόπου με του οποίου θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν κάποια προβλήματα σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Έτσι λοιπόν όπως όλοι γνωρίζουμε η Ένωση ήδη είχε την αρμοδιότητα να διαπραγματευτεί διάφορα ζητήματα σχετικά με τις επενδύσεις ακόμη και πριν τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας πιο σημαντικά η Ένωση ήδη μπορούσε να διαπραγματευτεί και έχει διαπραγματευτεί στοιχεία απελευθέρωση επενδύσεων. Αυτό που δεν έχει κάνει μέχρι σήμερα η Ένωση είναι να διαπραγματευτεί την προστασία των επενδύσεων μετά την εγκατάσταση. Αυτό ο τομέα παρέμενε στα χέρια των κρατών μελών και χρησιμοποίησαν ε, αυτή την αρμοδιότητα εκτατικά. Διαπραγματεύτηκαν πάνω από 1.200 ε, επενδυτικέ συνθήκε BATs, οι ε, περισσότερε ευρωπαϊκέ BATs Αυτές δηλαδή οι διμερείς συνθήκες επενδύσεω ακολουθούν ένα παρόμοιο μοντέλο, έχουν ευρύς ε, υποχρεώσεις ε, για το κέντρο υποδοχής ε, και τυπικά οι συνθήκες απαιτούν από το κέντρο υποδοχής να παράσχει εγγύηση στους ξένους επενδυτές συμπεριλαμβανομένες της εθνικής επιχείρησης, επιχείρησης του πλέον ευδομούνου κράτους κτλ. Επίσης απαιτούν από το κράτος υποδοχής να αποζημιώσει ένα ξένο επενδυτή σε περίπτωση απαλωτρίεση για να υπάρχει δίκαιη μεταχείριση και ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίου. Αυτές οι υποχρεώσεις τυπικά διατυπώνονται ε, με ιδιαίτερα ευρύ όρου και καθιστούν αδύνατο για τους επενδυτές και τα κράτη υποδοχής να προβλέψουν τις ε, αντίστοιχες υποχρεώσεις και τα δικαιώματα και η ασαφής διατύπωση που ακούσουμε έχει οδηγήσει τα δικαστήρια ε, να ε, έχουν εντελώς αντιφατικές ερμηνείες των ίδιων υποχρεώσεων. Το πιο διακριτικό χαρακτηριστικό στις συνθήκες ε, επενδυτικής προστασίας είναι ο μηχανισμός διευθυνσης διαφορών κράτους επενδυτή. Αυτό καθιστά τις ΜΕΙ διαφορετικές από οποιαδήποτε άλλη σύμβαση, ε, γιατί επιτρέπουν ε, στους ξενούς επενδυτές ε, να μηνύσουν το κράτος υποδοχής ενώπιον ενός πάνελ διαιτησίας, αν θεωρούν ότι έχει γίνει παραβίαση της συνθήκης. Οι επενδυτές μπορούν να προσβάλλουν ένα ευρύ μέτρο κυβερνητικών μέτρων σε μια τελική απόφαση διευθυνσίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τάσεις πριν από 15 χρόνια ε, δεν ε, ήταν ε, μια γνωστή διαδικασία αυτή η διατησία. Η πρώτη υπόθεση αποφασίστηκε το 1990, αλλά το 1994 μόνο, με την αυτά, μόνο στην αυτή περιλαμβανόταν ένα κεφάλαιο επενδυτικό και οι επενδυτές άρχισαν να χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο διευθέτησης διαφορών. Η πρώτη περίπτωση υπό την αυτά ήταν κατά του Καναδά, στην περίπτωση Εθήλ κατά του Καναδά. Ε, ε, ε, εκεί συμπεριλάμβανε μια νομοθεσία καναδική που απαγόρευε μια πρόσθετη ουσία βενζίνης για λόγους υγείας που ήταν ήδη απαγορευμένη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως αποτέλεσμα της διεκτησία, ο Καναδάς έκανε τρία πράγματα. Πλήρωσε την εταιρεία Ethel ζημίες για το κόστος και για, τα, για το διαφυγόν κέρδος κατέργησε την ε, νομοθεσία ε, περί υγείας και έκανε επίσημη δήλωση ότι η ουσία δεν έθετε κίνδυνο για την υγεία. Το προϊόν παραμένει ε, σε πάρα πολλέ άλλε δικαιοδοσίε απαγορευμένο από τότε. Έχουν υπάρξει 66 διευθετήσεις που κατατέθηκαν κατά τριών κρατών ναύτα, του Καναδά, τον ΗΠΑ και το Μεξικό και προσβάλλουν μια ευρεία σειρά μέτρων όπως περιβαλλοντικά μέτρα, περιβαλλοντικά μέτρα, μέτρα υγεία. Για αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία, ε, διαχείριση αποβλήτων και πολλούς άλλους τομείς. Τώρα μπορούμε να δούμε εδώ στο γράφημα ότι το κεφάλαιο 11 της ε, ΝΑΦΤΑ ήταν ε, ένα σημείο αφετηρίας για σημαντική αύξηση σε τέτοια επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτή και κράτους, όμως αυτό δεν περιοριζόταν μόνο στην ΝΑΦΤΑ. Ε, μπορούμε να δούμε ότι αυτή είναι η παγκόσμια τάση. Έχουμε περίπου 30 με 40 νέες τέτοιες διαδικασίες της ετησίως και αν το συγκρίνουμε αυτό με υποθέσεις στο ΔΕΚ ή στον ΠΟΕ, ο αριθμός ε, των υποθέσεων κράτους επενδυτή είναι πραγματικά εκπληκτικός ως προς το νούμερο και έχω βάλει εδώ ε, τις γνωστές ε, περιπτώσεις γιατί έχουμε και πάρα πολλές υποθέσεις που παραμένουν άγνωστες. Έτσι λοιπόν βλέπετε ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι γνωρίζουμε σαφήνεια τον αριθμό των υποθέσεων. Ε, αυτή η τάση εκδηλώθηκε και στην Ευρώπη. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης ε, είναι στόχοι ε, των ξενών επενδυτών υπό τις ε, συμφωνίες που έχουν υπογράψει. αναμένεται να υπάρξει και αύξηση στις υποθέσεις κατά της Ευρώπης στα χέρια του 2009, πάνω από 17% όλων των γνωστών διενέξεων επενδυτή κράτους ε, κατατέθηκαν κατά των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν ε, η Ευρώπη ε, έχει τέτοιες διευθυντήσεις με την Κίνα, την Ινδία, τον Καναδά και τις χώρες Μερκοσούρ μπορούμε να αναμένουμε ότι και αυτοί οι επενδυτές ιδίως δεδομένων των στρατηγικών που ακολουθεί η κινέζικη κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν αυτό τον κανονισμό διευθέτησης διαφορών. Εδώ μπορούμε να δούμε και πάλι τα ίδια αριθμητικά στοιχεία σε διαφορετικό φορμάτ. Τώρα, αν, παρούμε, α, αν δούμε με έναν διαφορετικό τρόπο την πολιτική επενδύσεων, τα γεγονότα μας λένε πάρα πολλά σημαντικά πράγματα. Καταρχήν, οι διενέξεις αυξάνονται ταχαίως, πολύ ταχύτερα από ε, ό,τι βλέπουμε σε οποιοδήποτε άλλο τομέα του Δημόσιου Διεθνούς Δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ο στόχος 62 γνωστών ε, τέτοιων αξιώσεων και τρίτον τώρα έχουμε ε, δεκαετή εμπειρία αλλά όχι μεγαλύτερη με τέτοια ε, διευθέτηση, διαιτησία μεταξύ κράτους και επενδυτή. Είχαμε πάρα πολλά αποκαλύφθηκαν ότι υπήρχαν πάρα πολλές ελλείψεις ε, στους ε, κανόνες και νομίζω ότι καθώς καταρτίζει τώρα υπό την πολιτική της Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα αυτό, καλό είναι να ε, δούμε ποια είναι τα προβλήματα που προέκυψαν από την εμπειρία μας και να τα επιλύσουμε. Τώρα, αν σκεφτούμε τις τάσεις που περιγράψαμε παραπάνω, ε, πρέπει να απομακρυνθούμε από τον τρόπο που σκεφτόμασταν ε, το 1959. Ε, τότε τα ευρωπαϊκά κράτη προσπαθούσαν να προστατεύσουν τις επενδύσεις τους σε αναπτυσσόμενες χώρες από την απαλωτρίωση και οι επενδυτικές ροές ήταν μονοδιευθυντικές σε μεγάλο βαθμό. Σήμερα ζούμε σε ένα πιο πολύπλοκο κόσμο και όπως ακούσαμε και από τη μελέτη LSC, e, και από την ανακοίνωση της ε, Κομισιόν του Ιουλίου η Ευρώπη θέλει να κερδίσει νέες αγορές ε, και ταυτόχρονα να δεχτεί και επενδύσεις από το εξωτερικό. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικές ε, οι σκέψεις αυτές καθώς διαπραγματεύεται η Ευρώπη τέτοιες επενδυτικές συνθήκες. Η Ευρώπη ως παραλήπτης επενδύσεων θα πρέπει να έχει κατά νου ότι θα μπορούσε να καταλήξει στο να υπερασπίζεται μια ευρύ σειρά νόμων νόμων και κανονισμών στα δικαστήρια. Έτσι λοιπόν ε, το πεδίο των μελλοντικών ε, συνθήκων θα πρέπει ε, να καταρτιστεί έχοντας αυτά κατά νου. Όταν είπα και ο Καναδά συνειδητοποίησαν ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο αυτών των ε, προς των μηνύσεων ε, έκαναν αμέσως ε, ερμηνείες, μάλλον έκαναν ερμηνευτικές δηλώσεις και προσπάθησαν να καθορίσουν πώς έπρεπε να μοιάζει η διαδικασία επίλυσης διαφορών. Έτσι λοιπόν διαφέρουν αυτές οι αυτοί οι μηχανισμοί σε σχέση με το τι έχουμε σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή μα τελειώνει ο χρόνο, νομίζω ότι πρέπει να μπούμε στην ουσία τη υπόθεση. Χρειαζόμαστε περισσότερη σαφήνεια και προβλεψιμότητα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την ε, απρόβλεπτη νομοθεσία που θα μπορούσε να εφαρμοστεί μέσω της επίλυσης διαφορών. Δεν έχω χρόνο να μπω σε λεπτομέρειες. Ε, όλα υπάρχουν ε, στην μελέτη του LSE, του London School of Economics. Δεν θα μπω εδώ λοιπόν στην ουσία, αλλά πριν να ολοκληρώσω θέλω να πω λίγα λόγια σε σχέση με τη διαδικασία διατησίας αυτή καθ' αυτή είναι το πιο ε, το πιο διακριτικό χαρακτηριστικό των ε, beats και το άλλο μέρος ε, μπορεί να προσβάλλει κυρίαρχες πράξεις. Ε, έτσι λοιπόν δίνονται αρμοδιότητες των δικαστηρίων στους ιδιωτικούς διαιτητές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί ότι θα συμπεριλάβει στις συνθήκες ε, της ε, διαδικασίας ε, προστασίας. Αν το κάνουμε αυτό, πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει διαφάνεια. Η Κομισιόν έχει δει ότι αυτό είναι πρώτη τη σημασία αλλά πρέπει και να διασφαλίσουμε ότι οι διαιτητές είναι αμερόληπτοι και ανεξάρτητοι. Σήμερα δεν ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί μπορούν να έχουν διαφορετικού ρόλους. Και τρίτον, πρέπει να διερευνήσουμε, μάλλον να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει έφεση, γιατί ε, δεν ε, μπορεί να υπάρχει ε, διόρθωση στο σημείο αυτό. και θα τελειώσω εδώ. Θέλω να πω ότι η Κομισιόν πρέπει να διασφαλίσει συνεκτικότητα με τι υπόλοιπε πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι αυτονόητο. Αλλά πρέπει να πω ότι αν ε, θέλετε να υπάρξει τέτοια εφαρμογή, αυτών των αρμοδιοτήτων θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα το πράξουμε. Ευχαριστώ πολύ. Αν κάποια θέματα δεν τα φίξατε, θα τα πείτε ίσως στις ερωτήσεις και απαντήσεις. Και τώρα ο καθηγητής Κρίστιαν Τίτιε από το Πανεπιστήμιο της Χάλε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στην ομιλία μου θα επικεντρωθώ σε δύο θέματα. Καταρχήν θα υπησέλθω σε κάποιες βάσεις του Διεθνούς Δικαίου το Προστασίας των Επενδύσεων και την ε, Διετησία σε αυτό το τομέα και μετά θα μιλήσω για την πρόταση κανονισμού και την ανακοίνωση της Κομισιόν. Η προστασία των ξένων επενδυτών μέσω διεθνούς δικαίου δεν είναι καινούριο φαινόμενο, αντίθετα ε, είναι ένας ρεαλιστικός τομέας που ανάγεται στην εποχή των χανζιαντικών 14 14ος-15ος αιώνας και παλιότερα και τώρα με πάνω από 2.700 διμερείς ε, συμφωνίες, BIT τα λέμε, ε, προστατεύονται και προωθούνται οι ξένες επενδύσεις. Καταρχήν αντιλαμβανόμεθα ότι οι ξένες επενδύσεις ε, εξαρτώνται από καλό πολιτικό κλίμα μεταξύ χώρας προέλευσης και ε, υποδοχής και δεύτερον οι επιχειρήσεις θέλουν νομική ασφάλεια Κατά κανόνα, σε ό,τι αφορά την απόσβεση και το κέρδος, έχουν μια διάρκεια οι ξένες επενδύσεις 10 με 20 χρόνια και μόνο αν ο ε, δυνητικός επενδυτής είναι σίγουρος ότι θα παραμείνει η οικονομική αξία της επένδυσης, μόνο τότε θα κάνει θα λάβει την επιχειρηματική απόφαση υπέρ της ε, ε, επέμβασης. Και αυτό χρειάζονται οι συμβάσεις. Ε, είναι δημοσίου δικαίου οι συμβάσεις ε, διότι ένα κράτος μόνο από το είναι διεθνούς δικαίου, συγγνώμη, μόνο το διεθνές δίκαιο μπορεί να είναι δεσμευτικό για το κράτος ενώ το εσωτερικό δίκαιο δεν επαρκεί αφού μπορεί το κράτος να αλλάξει την νομοθεσία του απλές συμφωνίες, συμβάσεις καλύτερα, contracts μεταξύ ενός επενδυτή και του εις χώρας υποδοχής δεν παρέχουν προστασία παρά μόνο λίγοι γιατί μια τέτοια συμφωνία δεν εμποδίζει το κράτος να αλλάξει το εσωτερικό του δίκαιο ώστε να μην αξίζει πια να μην έχει αξία η σύμβαση. Το 1959 υπογράφηκε η πρώτη διμερή συμφωνία για την, πρόθεση των επενδύσεων, την προστασία των επενδύσεων, ε, μια ε, ιδιωτική συμφωνία μεταξύ επενδυτή και χώρα υποδοχή μπορεί να διαμορφωθεί με τρόπο τέτοιο ώστε να υποχρεούται σε περίπτωση παραβίαση να αποζημιώσει το κράτο, αλλά μόνο οι πολυεθνικέ επιχειρήσει έχουν την οικονομική ισχύ να διαπραγματευτούν τέτοιε συμφωνίε με το κράτο υποδοχή. Όμως, οι διμερείς συμφωνίες διεθνούς δικαίου ε, καλύπτουν τα συμφέροντα όλων των οικονομικών υποκειμένων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσει. Αυτό ισχύει και για ρήτρε ε, που αφορούν την διαιτησία του ε, μεταξύ κράτους και επενδυτή. Πέρα από τη διπλωματική προστασία έχουν άμεσο δικαίωμα προσφυγής οι επενδυτές ε, το δίκαιο αυτό ε, δεν ε, υπόκειται σε πολιτικές αυθαιρεσίες έτσι, επειδή δεν υπάρχει εναλλακτική. Η ειδική διαιτησία είναι η μοναδική δυνατότητα ώστε να έχουν από κοινού την επί τη διαδικασία, οι επενδυτέ και τα κράτη. Γι' αυτό τα BIT, αυτές οι διμερείς συμφωνίες, είναι κεντρικό στοιχείο στο σύστημα των εγγύσεων για τις επενδύσεις που παρέχονται από πολλά κράτη-μέλη της Ένωσης αυτός ο κεντρικός μηχανισμός της προώθησης της ε, οικονομίας ε, ε, είναι δεδομένος όταν υπάρχει διμερή συμφωνία. Επίσης, πολλές φορές επικρίνεται το μπίτο ότι δηλαδή τα κράτη δεν έχουν πια policy space, ένα πολιτικό χώρο, δηλαδή δεν έχουν ρυθμιστικές ελευθερίες, αλλά δεν ισχύει αυτό γιατί οι περισσότερες διμερείς συμφωνίες δεν ρυθμίζουν την πρόσβαση στην αγορά. Το αν και κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα γίνει δεκτός ένας επενδυτής στο η χώρα υποδοχής, αυτό επαφίεται 100% στη διακριτική ευχέρεια του κράτους τα, ε, οι διμερείς συμφωνίες δεν εμποδίζουν στο να απορρίψει μια επένδυση ένα κράτος ή να επικαλεστεί θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή προστασίας του περιβάλλοντος. Η προστασία των εγκεκριμένων επενδύσεων μέσω των διμερών συμφωνιών ε, πάντοτε ε, η προστασία αυτή ε, βρίσκεται σε σχέση και ο νομοθέτης φροντίζει γι' αυτό και η διαιτησία ε, σε σχέση με την ανάγκη της προστασίας των δημοσίων γενικών συμφερόντων του κράτους. Αν υπήρξαν ε, ελάχιστες δύο μόνο βέβαια, όπου το κράτος καταδικάστηκε σε σχέση με μέτρα προστασίας. Είναι η υπόθεση Metal Clad και SD Myers. Ε, ήταν θέμα απαλωτρίωσης με βάση το άρθρο 1 του ε, πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάτι παρόμοιο και ε, καθαρά προστατευτικό μέτρο. Ε, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που είναι γνωστές και πρόσφατες μάλιστα, τα διαιτητικά δικαστήρια πάντοτε αναγνωρίζουν τα θεμητά κρατικά συμφέροντα για την προστασία του περιβάλλοντος και μάλιστα θυμίζω μια πρόσφατη απόφαση από Δευτέρα Αυγούστου 2010 στην Κεντούρα Corporation εναντίον του Καναδά που αφορούσε ρυθμιστικά μέτρα σχετικά με ένα ζυζανιοκτόνο όλες οι ε, ε, κατηγορίες ε, από την πλευρά του επενδυτή απερίφθησαν και ο τελευταίος καταδικάστηκε να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα και 2,8 εκατομμύρια για το κόστος των δικηγόρων στον Καναδά. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να... Ε, υπάρχει, ε, υπάρχει αυτή η δυνατότητα για την ε, αναβάθμιση της κοινωνικής ευημερία. Περνάω στο δεύτερο σημείο, την αρμοδιότητα της, Ευρω... της Κομισιόν. Η πρόταση του κανονισμού θεωρώ ότι νομικά πείθει, όμως θα μπορούσαμε να κάνουμε την κριτική ότι δεν διαφοροποιεί πρώτον μεταξύ των επιπτώσεων που θα έχει η μετάβαση αυτή αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τη συνδίκη της Λισαβόνας και θα επηρεάσει τα μπιτ των κρατών μελών καθ' αυτά. Δεύτερον, τι συγκεκριμένες δράσει των κρατών μελών μετά την 1η Δεκεμβρίου 2009 σε σχέση με τι τις συμφωνίε, συμφωνίες, τα BIT που έχουν και τρίτον, το ασύμβατο επιμέρου διατάξεων αυτών των BIT με το ε, δίκαιο τη Ένωση. Πρέπει καταρχήν να διαπιστώσουμε ότι η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, από μόνη της, μεμονωμένα δηλαδή, δεν επηρεάζει τα BIT των κρατών μελών, τα οποία από άποψη διεθνού δικαίου παραμένουν αμετάβλητα και σε, από άποψη δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν οι συμφωνίες νόμιμες και παραθέτω εδώ τον ε, Γενικό Εισαγγελέα Τιτσάν, ο οποίος διαπιστώνει ότι ε, η εξωτερική αρμοδιότητα ε, της κοινότητας σε τομείς που ρυθμίζονταν με συμφωνίες κρατών μελών δεν σημαίνει και δεν μπορεί να σημαίνει ότι αυτές οι συμφωνίες θα καταστούν ασύμβατες με τις διατάξεις και αρχές της διάκρισης των εξουσιών, των αρμοδιοτήτων. Ε, άρα λοιπόν, σε σχέση με τη μετάβαση αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ε, τίθεται θέμα άρθρου 2 παραγράφου 1 του, της νομο, σχετικής νομοθεσίας. Δεν χρειάζονται εξουδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα κράτη-μέλη για να διατηρήσουν τις συμφωνίες. στο κεφάλαιο 2 λοιπόν του σχεδίου κανονισμού της Κομισιόν θα μπορούσε να ε, διαγραφεί. Αυτό το σημείο όμως είναι σημαντικό, πολύ σημαντικό για λόγους νομική ασφάλειας. θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι τα BIT διμερεί συμφωνίε δεν επηρεάζονται από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Γνωρίζω μάλιστα μία περίπτωση όπου ένα τρίτο κράτος ε, αρνείται κεντρικές ε, νομικέ εγγυήσει σε έναν Ευρωπαίο επενδυτή. μετά την ε, συνθήκη της Λισαβόνας, ε, λέγοντας ότι ε, είναι, δεν ισχύει. Αυτό δείχνει τι ζημιά μπορεί να ε, υπάρξει εάν δεν ρυθμίζονται σωστά όλα αυτά τα θέματα. Επίσης, ε, είναι σαφές ότι σε περίπτωση αντίφασης ε, ε, συγκεκριμένης διάταξης ε, μιας διμερούς σύμβασης με το δίκαιο της Ένωσης, το κράτος μέλος υποχρεούται να ε, ρυθμίσει το θέμα και να μην υπάρχει πια το ασύμβατο. Αυτό το έχει πει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτή η κατάσταση που αναφέρθηκε και από τον συνάδελφο Γούλκοκ, ανταποκρίνεται ε, και σε παλιές συμφωνίες φιλίας, ναυσιπλοείας ή εμπορικές συμφωνίες των κρατών μελών. Ε, πέρα από το γεγονός ότι ε, πρόκειται για συμφωνίες που είχαν συναυθεί πριν από τη θέση ισχύ της συνθήκης της ΕΟΚ, η απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την, τον περιορισμό της έγκρισης αυτών των συμφωνιών ε, στηρίζεται στην, ε, σε μεμονωμένες διατάξεις που είναι ασύμβατες με τη συμφωνία. Κατά τα άλλα, οι παλιές συμφωνίες εξακολουθούν να ισχύουν. Ε, σε σχέση με Πρέπει να ισχύει λοιπόν το άρθρο 207 παράγραφος 6 της συνθήκης και οι γενικές διατάξεις περί του δημοσίου δικαίου. Υπάρχουν ορισμένοι προβληματικοί τομείς που θα πρέπει να ε, ρυθμιστούν μια ε, ε, νομικά συνεπής και οικονομικά υγιής επενδυτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάντα θα εξαρτάται από τα κράτη-μέλη λοιπόν, άρα είναι σημαντικό να έχουμε μικτές συμφωνίες. Ευχαριστώ. Thank you, um, let's move to the... Ευχαριστώ. Ας προχωρήσουμε και στον τελευταίο μιλητή, ο κύριος Φαντεχόφεν από το Business Europe. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και αξιότιμα μέλη αυτής της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σε αντίθεση με τους άλλους συγκεκριμένου ομιλητές εδώ, εγώ δεν είμαι νομικός, αλλά έχω συναντήσει πάρα πολλούς νομικούς όταν συζητούσαμε το θέμα αυτό. Αυτό δεν ξέρω τώρα είναι καλό ή κακό αλλά θα ε, πρότεινα να κρατήσουν ε, ε, στο χέρι τους τα πορτοφόλια τους κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης. Φυσικά αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα για την Business Europe. Οι επενδυτικές συμφωνίες είναι πάρα πολύ σημαντικές γιατί δίνουν το δικαίωμα να επενδύσει κανείς σε κλειστές αγορές και παράσχουν και παρέχουν προστασία στους επενδυτές σε χώρες όπου μπορεί να υπάρχει περιορισμένη προστασία από το νόμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, φυσικά ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής. Ε, ε, έτσι λοιπόν είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει την ελευθερία των επενδύσεων και να διασφαλίσει την ύπαρξη κράτου δικαίου για την προστασία των επενδυτών. Οι επενδύσεις είναι η ατμομηχανή της οικονομικής ανάπτυξης και φυσικά οι επενδύσεις μπορούν να συμβάλλουν στο να υπερβληθούν κάποια εμπόδια για το εμπόριο στο μέλλον. Επίση είναι πολύ σημαντικέ για πολλούς τους στόχους της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η ασφάλεια του εφοδιασμού, ο εφοδιασμός σε πρώτες ύλες, επενδύσεις ε, σε ε, έργα, ε, σε ορυχεία, project σε, στη Βόρεια Αφρική, κάποια άλλα project όπως ο Ναμπούκο για τον ενεργειακό εφοδιασμό. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει προστασία για να υπάρχει και κατάλληλη αποδόση των επενδύσεων. Όπως ξέρετε, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ ενεργές σε έργα υποδομών παγκοσμίω και πολλέ φορέ η απόδοση αυτών των επενδύσεων έρχεται μετά από 10-20 χρόνια και έχουμε συγκεκριμένου κανόνε και συμβάσει δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και χρειάζεται πάρα πολλέ φορέ νομική προστασία. Επίση, μα ανησυχεί στην Ευρώπη το θέμα τη προστασία τη τεχνολογία. Αυτό σχετίζεται με τι επενδύσει, ε, προστασία δικαιωμάτων πνευματική διοκτησία. Ε, ε, τα δικαιώματα αυτά πολλέ φορέ μπορούν να παραβιαστούν από του εμπορικού εταίρου που που προσπαθούν να επιβάλλουν την ε, μεταβίβαση τη τεχνολογική γνώση και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει κατά αυτού. Ευτυχώ οι Ευρωπαίοι επενδυτέ από τι μεγαλύτερε ε, ε, εταιρείε μέχρι και τι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει δεν λαμβάνουν παντού δίκαια μεταχειρήση όταν επενδύουν στο εξωτερικό και οι επενδυτικέ συμφωνίε παρέχουν ε, βασική ε, προστασία που εμεί θεωρούμε πολλέ φορέ δεδομένη εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό αφορά την ύπαρξη ασφάλεια δικαίου. Κάτι που λείπει πολλέ φορέ σε αυτέ τι χώρε. Έχουμε κάποιε αλλαγέ κατόπιν τη θέσεω ισχύ τη συνθήκη τη Εμεί Εμείς υποστηρίζουμε αυτή την ενσωμάτωση στην εμπορική πολιτική γιατί είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσει κοινού κανόνε ε, για ε, το στάδιο πριν αλλά και μετά την εγκατάσταση εξάρτητα από τη χώρα καταγωγής. Και εμεί πιστεύουμε ότι αυτό θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, διαπραγματευτεί πιο φιλόδοξε συμφωνίε με τους εταίρους. Εμείς χαιρόμαστε που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέλεξε να μελετήσει αυτό το πολύπλοκο θέμα μέσω τη μελέτη του London School of Economics αλλά και με τη σημερινή ακρόαση σε ό,τι αφορά το σχέδιο του κανονισμού για την έγκριση ε, και για τον κανονισμό grandfathering. Ε, το Business Europe υποστηρίζει αυτό το σχέδιο κανονισμού αν θερμά γιατί θέλουμε να παράσχουμε το μέγιστη ασφάλεια δικαίου ε, για του επενδυτέ που έχουν επενδύσει στα κράτη-μέλη μέσω των BITs. Και φυσικά αυτό είναι και ο στόχος του κανονισμού. Σε ό,τι αφορά το grandfathering έχουμε μία ερώτηση. Θέλουμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς οι ρήτρε αναθεώρηση θα λειτουργήσουν στην πράξη για να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα μότρα με κανένα τρόπο δεν θα απειλήσουν ε, κάποιες εταιρείες ή επενδυτές που είναι τώρα σε διαδικασία ε, διατησίας με τρίτες χώρες. Επίσης, ε, θέλουμε να δούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαπραγματευτεί ευρεία συμφωνίες προστασίας ε, βάση της ε, πρακτικής που έχουν τα, ίδια τα κράτη-μέλη παρά να δουμε η ευρωπαικη ενωση να διαπραγματευτει ευρεια συμφωνιες προστασιας ε βασει της πρακτικης που εχουν τα κρατη μελη παρα να ξεκινησει απο το μηδέν. Έτσι λοιπόν, ε, δεν είμαστε σίγουροι ότι ο μηχανισμός όπως περιγράφεται στο σχέδιο κανονισμού είναι ο ορθός μηχανισμός, αλλά είμαστε ανοιχτοί στο να το συζητήσουμε αυτό και με τους λοιπούς πρωταγωνιστές. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω την αναθεώρηση των BATs σε σχέση με το αν συνάδουν με τις συνθήκες για τη μεταφορά κεφαλαίου. Κατανοούμε ότι υπάρχουν ε, πρακτικές συνέπειες για τις πολιτικές της Ένωσης σε σχέση με τους ε, χρηματοοικονομικούς περιορισμούς για χώρες όπως το Ιράν και άλλες, αλλά οι θεσμοί τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να γνωρίζουν ότι και η μεταφορά κεφαλαίου είναι σημαντικό θέμα για την ασφάλεια των επενδύσεων και αντιμετωπίζουν οι εταιρείε μας τέτοιο ε, πρόβλημα καθώς αποσύρονται από το Ιράν λόγου χάρη σε ό,τι αφορά το empowerment. Πιστεύουμε ότι αυτή είναι μια θετική πτυχή του κανονισμού, αν και είναι δύσκολο για μας να δούμε πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Και φυσικά δεν θα έπρεπε αυτό να φρενάρει την ανάπτυξη μιας ε, πολιτικής επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα θα στραφώ στις μελλοντικέ επενδυτικέ πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ανακοίνωση. Πιστεύουμε ότι η ανακοίνωση της Κομισιόν παρουσιάζει ε, τα σχετικά θέματα για τις επιχειρήσεις ε, πρώτη εγκατάσταση ή για την πρόσβαση στην αγορά. Η ανακοίνωση βασικά βασίζεται στην τρέχουσα πρακτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που βασίζεται ε, στι υπηρεσίε Θεωρούμε ότι αυτό θα πρέπει να έχει συνεχιστεί και να υπάρχει ευρύτερη κάλυψη για την ε, βιομηχανία και για ε, τις υπηρεσίες και για τι σχετικέ συμφωνίε στο μέλλον. Ε, σε ό,τι αφορά το στοιχείο μετά τις εγκατάστασεις για την προστασία των επενδυτών, δηλαδή θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει ε, εις ε, την πρακτική που ακολουθείται στα κράτη-μέλη στα, πλαίσια των BIT και θέλουμε να υπάρχουν σημαντικέ αρχέ όπω μη διάκριση, ε, εθνική μεταχείριση προστασία κατά της απαλωτρίωσης, οι λεγόμενες ε, ρήτρε ομπρέλα, γιατί πιστεύουμε ότι από την επιχειρησή σκοπιά αυτές οι αρχές επεκτείνουν την ερμηνεία της Ένωσης του κράτους δικαίου για την προστασία των επενδυτών σε χώρες όπου τα νομικά του συστήματα είναι λιγότερο ανεξάρτητα και δεν λειτουργούν τόσο καλά όπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δυστυχώς υπάρχει και κακοδιαχείριση. Επίσης, ε, θα ήθελα να αναφερθώ στην ε, μελέτη του London School of Economics. Υπάρχει ένα σημείο βέβαια που προκαλεί κάποια σύγχυση. Δεν πρέπει να υπάρχει σύγχυση μεταξύ της πρόσβασης στην αγορά για τους επενδυτές και της προστασίας των επενδυτών η πρόσβαση σε συμφωνίε ε, πρώτη εγκατάσταση συχνά περιλαμβάνει περιορισμού. Παραδείγματο χάρη, μια χώρα που έχει του πόρου πολλέ φορέ θα αποκλείσει του φυσικού πόρου γιατί θα θεωρήσει ότι είναι στρατηγική σημασία για την οικονομία. Έτσι λοιπόν μπορεί να μην υπάρξει πρόσβαση στην αγορά για αυτού του πόρους, αλλά μπορεί να είναι αποδεκτό να επιτρέψει εξαίρεση για την προστασία των επενδυτών από αυτό το τομέα, γιατί θα μπορούσε αυτή η χώρα να καλέσει νέου επενδυτέ, να συμμετάσχουν σε ένα πετρελαϊκό έργο, παραδείγματο χάρη, όπου θα χρειαστούν μεγάλε επενδύσει και θα χρειαστεί αυτό ο επενδυτή πλήρη προστασία. Αυτό είναι σημαντικό θέμα λοιπόν. Ξέρω ότι έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις ε, για το αποκαλούμενο public policy space και το αρνητικό αποτέλεσμα των επενδυτικών συμφωνιών. Η Business Europe διαφωνεί με αυτό το επιχείρημα ότι οι επενδυτικές συμφωνίες θα υποσκάψουν τους περιβαλλοντικούς ή τους ε, κοινωνικούς ε, κανόνες, τη σχετική νομοθεσία, γιατί η νομολογία δεν υποστηρίζει την άποψη αυτή, γιατί οι διαιτητές εφαρμόζουν κανόνες αναλογικότητας, όπως θα, ήταν, θα ίσχυε και σε εγχώριες υποθέσεις Νομίζω ότι πολλές αποφάσεις ε, επιτρέπουν ε, στις κυβερνήσεις να ρυθμίσουν και επίσης ε, θέλω να πω ότι κρατημέλη είναι μέρη στις περισσότερες σε όλο τον κόσμο και παρόλα αυτά δεν υπάρχει ένα τέτοιο regulatory chill στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλα αυτά έχουμε τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα σε όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν λοιπόν, αν κάποιο θέλει να ε, μου εξετάσει εμένα αυτό τον αρνητικό αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα τον ευγνωμονούσα. Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ ότι πολύ συχνά σε μεγάλες ε, επενδυτικές υποθέσεις εμπλέκονται και ε, οι κυβερνήσεις. Ε, πολλές φορές χρησιμοποιούνται κανόνες για την υγεία των περιβάλλων ή τη φορολογία για να γίνει μια απολωτρίωση. Πολλές εταιρείες έχουν κατηγορηθεί αδίκως ότι παραβιάζουν αυτή την νομοθεσία λόγω μιας ε, απόφασης ε, διαιτησίας όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν θα πρέπει να υποχωρήσει προς αυτά τα κράτη που προσπαθούν να κλέψουν την τεχνολογία και τις επενδύσεις μας. Αν δούμε τις κατευθυντήριες CSR εκεί υπάρχουν παρόμοιοι κίνδυνοι από τις χώρες που υιοθετούν παράτυπες πολιτικές. Τώρα, πιστεύουμε ότι ίσω για αυτέ τι κατευθυντήριε γραμμέ, ε, CSIR μπορεί να μην είναι καλό να τι συμπεριλάβουμε στι μελλοντικέ συμφωνίε. Ε, δεν ε, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα εφαρμογή αυτών των κατευθυντήριων γραμμών ε, στι ευρωπαϊκέ εταιρείε, γιατί τίνουν οι ευρωπαϊκέ εταιρείε να εφαρμόζουν αυτέ τι κατευθυντήριε γραμμέ και υπάρχει ένα δίκτυο κανόνων που πρέπει να σεβαστούν οι ευρωπαϊκέ εταιρείε. Υπάρχουν και μηχανισμοί στα κρατη μελη και στον ΩΣΑ που λειτουργούν αποτελεσματικά. Οι ανταγωνιστέ μα από τι ε, χώρε όπω ε, Κίνα και Ρωσία δεν πρέπει να ακολουθήσουν αυτέ τι κατευθυντήρες γραμμέ, και αυτό είναι το κύριο πρόβλημά μα, και θα προτιμούσαμε να έχουμε μια νέα στρατηγική προκειμένου αυτέ οι αναδυόμενε οικονομίε να προσυπογράψουν αυτέ τι κατευθυντήρες γραμμέ, έτσι ώστε να έχουμε του ίδιου κανόνε για όλου όσου λειτουργούν στην παγκοσμία αγορά. Τέλος, ε, σε ό,τι αφορά την επιλύση των διαφορών και τη διατησία, υποστηρίζουμε τις προτάσεις στην ανακοίνωση να χρησιμοποιήσουμε ε, μηχανισμούς ε, κράτους προκάτους και μηχανισμούς διευθέτησης επενδυτή κράτους. Δεν μπορούμε να, συμφωνούμε, να συμφωνήσουμε με το ότι αναφέρεται ότι δίνονται ειδικά δικαιώματα στις επιχειρήσεις. Εδώ ε, πολλές φορές πρέπει να εξετάσουμε τι γίνεται με το κράτος δικαίου, αν είναι αδύναμο. Υπάρχει και ένα θέμα για τα πάνελ της διαιτησίας βλέπουμε πρόβλημα, είναι το υψηλό κόστος αυτών των πάνελ και αυτό είναι δύσκολο να το καλύψουν οι μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Μπορούν να υπάρξουν μέτρα για να, ε, να χορηγούν χρηματοδότηση στις ΜΜΕ για να χρησιμοποιούν αυτούς τους μηχανισμούς ή να ε, δίνονται περισσότερες εγγύσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Σας ευχαριστώ. Uh, Έχουμε τελειώσει με τις τρεις παρουσιάσεις. The Business uh, Association. Uh, let's move to the... Περάσουμε τώρα στα μέλη της Επιτροπής, αρχίζοντας ε, με τον εισηγητή, τον Κάλσιτα από τους Πράσινους, που ήταν εισηγητής για την ε, για τον κανονισμό όταν έγινε η συζήτηση του, της μεταβατικής περίοδου προς τον κανονισμό. Και επίσης ε, θα περάσουμε ε, μετά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, μπορούμε να σας ακούσουμε, θέλετε να μας πείτε τις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις σας και τους τρεις και ευχαριστώ Γλυκό για την έκθεση που μας υπέβαλες. Θα ήταν ε, πολύ βοηθητικό για μας, τονίζω, και θα ήταν και πάρα πολύ χρήσιμο για την εργασία μας να υπήρχε αυτό το κείμενο στη διάθεσή μας. Όταν το διαβάζω βλέπω ότι τίθενται μερικά ερωτήματα. Ε, θα ήθελα να σας τα θέσω και υπάρχει και το θέμα των διαπραγματεύσεων που θα έπρεπε να είναι στο επίπεδο των διεκδικήσεων των κρατών μελών που έχουν αναπτύξει τα πράγματα όπως λέγεται και στα συμπεράσματα. Ποιο είναι το συμπέρασμα τελικά, θέλουμε αυξημένη προστασία ως προς το, την έμεση απαλωτρίαση θα έχουμε ε, προσθήκη της ε, ε, αναπτυξιακής πηγής. Μας μιλάτε για τις διάφορες επιπτώσεις και για τη διαχείρισή τους, αλλά δεν είναι αρκετά. Δεν ξέρω αν είναι μέσα στα καθήκοντά σας να τα προσδιορίσετε πιο ακριβώς όλα αυτά. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι μια πιο ακριβής διατύπωση και επίσης για τις εναλλακτικές λύσεις, των, για τις εναλλακτικές πολιτικές που υπάρχουν, ε, θα θέλαμε να ξέρουμε πώς θα πρέπει να αντιδράσουμε στις ε, ερωτήσεις που θα θέσουμε για τον κανονισμό. αυτά τα έγραψα και δεν τα ξεχνώ. Τώρα, μιλάτε για την συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία αφήνει ανοιχτές μερικές προδιαγραφές, την ανάπτυξη των πολιτικών, ε, ότι θα πρέπει να μην υπάρχει επικάλυψη, θα πρέπει να την αποφεύγουν τα θεσμικά όργανα και δεν νομίζω ότι το επιτρέπει αυτό να γίνει η συνθήκη της Λισαβόνας. Υπάρχει ένας κανόνας ε, ε, που προσδιορίζεται από την οδηγία, την υπάρχουσα. Τώρα πώς θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε τα κράτη-μέλη από το μποϊκοτάρισμα της ε, πολιτικής της ΕΕ. Τι πρέπει να αλλάξει εδώ για να υπάρχει αποτελεσματικότητα. Και επίσης υπάρχει η μεταρρύθμιση της πολιτικής αυτής. Πριν να έχω μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική έχουμε τον ΠΟΕ. Αλλά βεβαίως όλα αυτά είναι χρονοβόρα, η διαδικασία θα κρατήσει καιρό και συνεπώς εάν θέλετε να υπάρχει μία λύση μέσα σε ένα έφθετο χρονικό διάστημα στον τομέα του εμπορίου πρέπει να γίνουν διαπραγματεύσεις. Τι βλέπετε λοιπόν ως επιλογές πολιτικής στο έγγραφο της ε, Επιτροπής που υπάρχει δυνατότητα να αποσυρθούν, υπάρχει η δική σας πρόκληση των νέων προτάσεων και υπάρχουν και οι παλιές. Γιατί μία από τις επικρίσεις μου για το σχέδιο κανονισμού είναι σε ένα άρθρο λέει ο μιλητής το 6 έχει ε, αποσυρθεί και το 5 έχει αλλάξει. Ε, είναι να υπάρξει μια αποσαφήνιση στο τελευταίο άρθρο είναι, υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον να αρθούν τα εμπόδια για τις ε, ε επενδύσεις στην ΕΕ. Νομίζω όμως ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Έχουμε και άλλους στόχους, πάρα πολλούς και ποιε θα ήταν οι επιπτώσεις όταν προσθέτουμε και άλλα πράγματα στο σημείο αυτό. Ή ας πούμε η αηφόρος ανάπτυξη, ε, η συμπερίληψη προβλέψεων διαρκούς ανάπτυξης, ε, πώς θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να επαναδιαπραγματευτούν αυτούς τους όρους, αν θέλαμε να τους εισάγουμε και μετά η νομική αβεβαιότητα. Νομίζω ήταν σημαντικό ε, το ότι προτείνατε ορισμένα μέτρα ως προς τη νομική αβεβαιότητα διότι από τη στιγμή ότι αυτά, που αυτά τα κείμενα δεν έχουν ε, ε, νομική ισχύ, δεν βασίζονται μόνο στη συνθήκη έχουν μια νομική βεβαιότητα όχι επειδή προέρχονται από ένα δικαστήριο αλλά έχουν μια νομιμότητα επειδή βασίζονται στη συνθήκη. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε ότι δεν έχουμε δυνατότητες ε, παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, υπάρχει μια γενικά ε, ασάφεια ως προς το σημείο αυτό, μια νομική αβεβαιότητα. Νομίζω ότι θα πρέπει να καταρτήσετε μια σειρά κριτηρίων, ούτω ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ε, να υπάρχει ένα νομικό φάσμα υποχρεώσεων και να κάνει μια αξιολόγηση του η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να δει ότι αυτή η συμφωνία συμφωνεί με τους κανόνες και την οδηγία και συμφωνεί, καλύπτεται από τη συνθήκη και τότε αισθάνομαι πολύ καλύτερα και λέω ότι έχουμε ακολουθήσει την κανονική διαδικασία Κανεί δεν λέει παραδείγματο χάρη ότι καταργώντα το κεφάλαιο, διαγράφοντας το κεφάλαιο 2 έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι κανεί μπορεί να θέσει ένα αμφιβόλο την νομιμότητα αυτού του κειμένου που καλύπτεται από τι συνθήσει. Θα ήθελα να ακούσω τα σχόλιά σας πάνω στη μακρά δήλωση που μόλι υπέβαλα και μετά θα ήθελα να στραφώ προ την Αταλή δεν μπορώ να, να προφέρω καλά τα άλλα δύο ονόματά σας, Ναταλή, γι' αυτό. Νομίζω ότι μιλάτε για κάτι πολύ ενδιαφέρον καταρχήν, θίγεται ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Το θέμα της επίλυσης διαφορών. Πολλοί συνάδελφοι το τόνισαν αυτό και έχει σχέση με τη διαφάνεια γιατί σύμφωνα με την ε, συνθήκη της Λισαβόνας και δίνει πρόσβαση στις τρίτες πλευρές, στα τρίτα μέρη, δηλαδή τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και τα λοιπά. Πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και πώς, εάν ναι, να υπάρχει ένα άνοιγμα. I'll finish this question soon, but ε, Υπάρχουν και άλλα ερωτήματα που θα ήθελα να θέσω στη σειρά στη συνέχεια αναφέρατε, εσείς το είπατε, ότι έχουμε μία νομολογία η οποία λέει ότι δεν υπάρχει νομικό εργαλείο. Δεν ξέρω, εδώ έχει υπάρχει μια αντίφαση για μένα, δεν το ε, καταλαβαίνω αυτό παρά μόνο αντιφατικά. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω να υπάρχει μια κοινή δημόσια γνώμη, ε, βάση με συγχωρείτε δεδομένων, και θα ήθελα να υπάρχει ένα κανονικό δικαστήριο που να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται, για ποια θέματα μπορούμε να προσφύγουμε σε αυτό το δικαστήριο και συγκεκριμένους δικαστές αυτό θα ήταν ε, το σωστό για μένα και όχι να έχουμε όλα τα διαιτητικά δικαστήρια, άγνωστους ανθρώπους και άγνωστα δικαστήρια που να ασχολούνται με όλα αυτά τα θέματα. Επίσης, πέστε μου για την ε, βάση δεδομένων, τη διαθεσιμότητά της, ε, τις δυνατότητες παρέμβασης, την πρόσβαση κτλ και θα ακούσω τις απαντήσεις και ελπίζω να επανέλθω μετά γιατί θα έχω και άλλες ερωτήσεις άμα ρωτάτε τόσο πολύ, δεν θα έχουν χρόνο να σας απαντήσουν. Ευχαριστώ πολύ, ε, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους τέσσερις ε, παρεμβαίνοντες για την ποιότητα των ανακοινώσεών τους. Πιο δυνατά λέει το ακροατήριο την ποιότητα λοιπόν των ανακοινώσεων τους και μας έδωσαν ε, μια τεχνογνωσία που είναι δική τους για ένα θέμα πάρα πολύ δύσκολο που οποιοδήποτε βουλευτής πρέπει να, να δεχτεί ότι δεν το γνωρίζει πολύ καλά. Εγώ είμαι σκιώδης εισηγητής ε, στο θέμα που ανάφερε ο κύριος Ντερ και επίσης ε, είμαι και εισηγητής στο θέμα ε, με το, σύμφωνα με το οποίο συνάντησα όλους τους άλλους εκπροσώπους, της μη κυβερνητικέ οργανώσεις, για να καταλήξω σε μια εργασία η οποία θα πρέπει να περατωθεί κανονικά τον επόμενο Μάρτιο και θα γίνει μια ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Απριλίου. Οπότε καθ' όλη αυτή την περίοδο θα υπάρχει συζήτηση με τους διάφορους εταίρους. Η προτεραιότητά μου είναι να στραφούμε σε πέντε κεφάλαια το πρώτο μου κείμενο που αφορά τον ορισμό και το πεδίο εφαρμογής ε, για τις ε, επενδύσεις, το δεύτερο κεφάλαιο η προστασία των επενδυτών, το τρίτο ε, η προστασία του κοινού και ο μηχανισμός του, της επιλύσεως διαφορών και η διεθνής ευθύνη η διευθύνη μάλλον σε διεθνές επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή εγώ ήμουν εισηγητής για την πολιτική των επενδύσεων, πρέπει να πω ότι το Κοινοβούλιο θα έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει από αυτού. Για μένα είναι προτεραιότητα, γιατί ε, αντικατοπτρίζει πάρα πολύ σωστά το κοινοτικό συμφέρον. Είναι ένας δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε, που τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι θα ανήκει κανονικά στην, ε, στον ιδιωτικό τομέα. Για μένα είναι το πρώτο θέμα, ο χώρος παρέμβασης του, ε, για το δημόσιο. Νομίζω ότι πρέπει να διαλέξουμε καταρχήν τις ομάδες και να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν ορισμένες αρχές. Σημαντικό θέμα είναι και οι διαπραγματεύσεις των ΩΣΑ που είχαν ε, ε, βαρύνει στην ε, ε, Επιτροπή των Επενδύσεων και ε, η οποία είχε ασχοληθεί με θέματα που όλα αφορούν τον Ευρωπαίο πολίτη της αύριο. Ας ρωτήσουμε λοιπόν αν μπορούμε να αφήσουμε μια ιδιωτική επιχείρηση να επιτεθεί μια κυβέρνηση για την κοινωνική ή την περιβαλλοντική της πολιτική. Αν μπορούμε να αφήσουμε έναν επενδυτή να κερδίσει τη δυνατότητα της έφεσης χωρίς να υπάρχει διαφάνεια ε, στην ετοιμιγορία ούτε στο περιεχόμενο ε, και οπότε ε, θα γίνει μια πληρωμή σύμφωνα με ποια κριτήρια. Δεχόμαστε οι μεγάλες επιχειρήσεις να γίνονται δεκτές σε μεγάλες αγορές όπως είναι της Κίνας ή της Ινδίας όταν δεν είναι και τα δυο μαζί όταν αρχίζουν με ε, ξένες επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς. Το παράδειγμα του πυρηνικού τομέα, η συνεργασία με την Κίνα, το θέμα της κουλτούρας, το θέμα της παιδείας, εκπαίδευσης. Θα δεχτούμε να υπάρξει μια ενισχυμένη προστασία των ξένων επενδύσεων, ε, η διαχείριση των ε, πορτφόλιων την, ε, σε σχέση με την Κίνα η οποία έχει τεράστιες δυνατότητες σε αυτό το τομέα, η προστασία των επιχειρήσεων γιατί και αυτές κάνουν επιθετικές επενδύσεις, έχουμε τη δυνατότητα να τις προστατέψουμε. Όλες αυτές τις ερωτήσεις τις θέτω στον εαυτό μου καταρχήν και θα τις βρούμε στο δικό μου το κείμενο, είναι γραμμένες μέσα θα ήθελα να περατώσω θέτοντας δύο ερωτήματα στους παρεμβαίνοντας, τους δύο από αυτούς τουλάχιστον. Ε, στον κύριο Γουτκοκ θα ήθελα να ρωτήσω για τις ε, μελλοντικές συμφωνίες επενδύσεων της Ευρώπης θα πρέπει να φτάνουμε σε ποιο βαθμό ε, ευκρίνειας και για την κυρία Ρεσπόνη θα πρέπει να ρωτήσουμε την κυρία Μπερνασκόνη για τις ε, δυνατότητες αντιμετώπισης ξένων επιθέσεων ε, και έχουμε ορισμένα πρότυπα τα οποία τα ανάφερε πριν από λίγο ε, το καναδέζικο μοντέλο και το αμερικανικό είναι πρότυπα αυτά τα δύο για την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ας ανοίξουμε τώρα τη συζήτηση και στα άλλα μέλη της Επιτροπής. Λοιπόν, πρέπει να βάλουμε ένα όριο στο χρόνο ομίλιας. Επίσης, ε, οι ακροάσεις σκοπό έχουν να μας επιτρέψουν να ακούμε τους προσκεκλημένους, όχι τον εαυτό μας. Μίχελ, από την ομάδα των φιλελευθέρων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχήν να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες για τις ομιλίες τους που μας έδωσαν σημαντικές ε, γνώσεις. Συμπληρωματική ερώτηση παρακαλώ. Η συζήτηση εδώ κινείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ένα πεδίο έντασης υπάρχουν διαφορές μεταξύ κρατών μελών ανάλογα από το αν υπάρχουν ή όχι ε, και αν υπάρχουν πώς έχουν διαμορφωθεί. Τα κράτη και οι επενδυτές, οι επιχειρήσεις που έχουν συνάψει ε, ικανοποιητικές συμφωνίες δεν θέλουν να τις αλλάξουν. Αυτό είναι σαφές. Τώρα, από τεχνικής πλευράς, τι γίνεται, ποια διαδικασία θα βρεθεί, ώστε και οι άλλες χώρες να πάρουν ένα τέτοιο υπόδειγμα συμφωνίας. Ίσως ο καθηγητής Τίτια μπορεί να μας πει. Δηλαδή, μπορεί να υπάρξει κάποια κοινοτικοποίηση, ας πούμε, με την έννοια του κοινοτικού συντονισμού, ώστε να ε, υπάρξει ας πούμε μια τέτοια νομική ε, δυνατότητα. Ο συνάδελφός μου μίλησε πολύ πιο λίγο από ό,τι φανταζόμουν, γι' αυτό δεν ήμουν στο έδρανό μου. Στην ε, έκθεση περίληψη λέει ότι οι προτινόμενες εξουσίες για την Κομισιόν για να αποσύρει την έγκριση το, στα ε, θα προσθέσει και δεν θα μειώσει την νομική ασφάλεια. Αλήθεια είναι αυτό. Και λίγα λέμε όχι. Ε, ε, ε, αυτό δεν, δεν είναι σωστό. Εδώ νομίζω ότι υπάρχει μια απειλή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε εσωτερικές επενδύσεις περισσότερες από τον καθένα για πολλά χρόνια. Το 60% στις τελευταίες ευρωεκλογές ψήφισαν κατά τις συνθήκες της Λισαβόνας και με αυτό τώρα απειλείται η ικανότητά μας να είμαστε ανταγωνιστικοί σήμερα. 400 θέσεις εργασίας χάθηκαν σήμερα στο, στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από με την κατάσταση στην Πολωνία. Δεν έχω, τη συμπαθώ τη χώρα, αλλά ε, εδώ έπαιξαν ρόλο οι επιδοτήσεις. Τώρα απειλείται και η ε, η δυνατότητα που έχουμε να πάρουμε πίσω αυτές τις θέσει εργασίας λόγω ακριβώς των ε, συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών. Επανέρχω, πριν να δώσω το λόγο στην Επιτροπή, πριν δώσω το λόγο στους προσκεκλημένους μας. Ο κύριος Πετριτσόνε. Η Κομισιόν λοιπόν θα μας πει τη γνώμη της. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε η ακρόαση αυτή αφορά κυρίως τους εμπειρογνώμονες που πρέπει να τους ακούσουμε. Τέσσερις σύντομε παρατηρήσεις για να θυμίσω το πνεύμα της Κομισιόν όταν υπέβαλε το αυτό το πακέτο. Πρώτον, νομίζω το είπαν και πολλοί, και κάποια μέλη της Επιτροπής. Αυτή η αρμοδιότητα είναι καινούρια, αλλά έχει παρελθόν. Το πνεύμα του πακέτου είναι να προσθέσει και όχι να αφαιρέσει αξία από την υπάρχουσα κατάσταση. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα ως συνέπεια. Πρώτον, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ε, ευρωπαϊκών ενωσιακών μπιτ και των ε, εθνικών μπιτ. Ε, τα κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης θα βελτιώνουν ή όχι την κατάσταση. Αυτό θα πρέπει να δούμε. Μην ε, ε, υπερτονίζομαι το θέμα των αρμοδιοτήτων. Όλα τα θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη ε, είναι υπέρ των αρμοδιοτήτων. Πολλές φορές όμως το παρακάνουμε, παρασυρώμεθα. Εμείς κάναμε μια επενδυτική πολιτική σε συμφωνία με τα κράτη-μέλη, εξελίχθηκε αυτή παρά το θέμα της αρμοδιότητας και η προσέγγιση της Κομισιόν να συνεχίσουμε αυτή την εξελικτική πορεία σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη. Δεύτερη παρατήρηση. Πρόκειται για μεταβατική φάση τώρα. Πάλι αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να διαιωνίζουμε την υπάρχουσα κατάσταση. Πρέπει κάποια στιγμή να γίνει κάτι που θα σηματοδοτεί ότι ο κόσμος των beach έχει αλλάξει. Παράλληλα, όλοι συμφωνούν ότι η ανατροπή της υπάρχουσας κατάστασης σε μια νυχτή θα ήταν καταστροφική. Η ρήτρα επανεξέταση είναι προσπάθεια Κομισιόν να βρει μια ισορροπία μεταξύ των δύο άκρων. Δεν, έχουμε, δεν μονοπολούμε τη σοφία, ούτε είναι η μόνη μέθοδος για να βρεθεί μια ισορροπία. Κάναμε μια συζήτηση στους κόλπους της Κομισιόν, χωρίς να συμφωνήσουμε όλοι υπέρ της καλύτερης μεθόδου. Αλλά ε, το βασικό είναι ότι χρειάζεται μια ισορροπία που θα δείχνει ότι η φυστάμενη κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί αενάως και από την άλλη δεν μπορεί να ανατραπεί ε, ξαφνικά. Τώρα για το θέμα των διαφορών. Δεν εκπλήσει ότι υπάρχουν ε, διαφορές α, ε, απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία διευρύνθηκε πολύ και είναι ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής. Και αν δούμε την αναλογία των 60 περίπου υποθέσεων ε, γενικά και αν δούμε ε, την Ευρώπη και τις επενδύσεις ε, θα δούμε ότι είναι λιγότερες οι προβληματικές υποθέσεις και διενέξεις που έχουμε. Δεν σημαίνει ότι η επίλυση των διαφορών δεν είναι θέμα, είναι θεμελιώδες μάλιστα, αλλά θα πρέπει να έχουμε ουσιαστικά πρότυπα σημαντικά, ουσιαστικού δικαίου και θα πρέπει να έχουμε και τις σωστές διαδικασίες. Μιλήσαμε για τη διαφάνεια, υπάρχουν και άλλα θέματα που πρέπει να δούμε εδώ η Κομισιόν έχει καταδείξει ορισμένα, υπάρχουν και άλλα. Τέλος. Γιατί υπάρχει στη συνθήκη επενδυτική πολιτική. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αντιμετωπίζει καλά με βάση τα παγκόσμια πρότυπα τον ε, ξένο επενδυτή. Θέλουμε οι ξένοι επενδυτές μας να έχουν μεταχείριση παρόμοια με αυτή που έχουμε στην Ευρώπη. Οι ξένοι επενδυτές θα έχουν μια διασφάλιση ότι θα συνεχίσουμε να τους παρέχουμε τη μεταχείριση που προβλέπουν οι νόμοι μας. Αυτό είναι ε, το βασικό. Ο στόχος οι τεχνικές λεπτομέρειες μπορεί να είναι ε, ε, διαβολικά περίπλοκες, αλλά το κριτήριο συγκριτικής αξιολόγησης, το benchmark, είναι να δούμε τι κάνουμε εμείς στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις και να επιτύχουμε ένα παρόμοιο καθεστώς για τους δικούς μας επενδυτές που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Ευχαριστώ. Ας επανέλθουμε με την ίδια σειρά στους καλεσμένους μας. Θα δώσω το λόγο καταρχήν στον καθηγητή Ούλκοκ. Πρέπει να περιοριστείτε στα πέντε λεπτά. Ο καθένα θα πρέπει να περιοριστεί στα πέντε λεπτά. Κύριο Γουλκοκ, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ και για τι ερωτήσει που θέσατε. Θα προσπαθήσω να τι καλύψω όσο καλύτερα γίνεται δεδομένου του χρόνου σε σχέση με το ε, πρέπει να ε, συντεριάξουμε τις ε, beats των κρατών μελών. Αν οι διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συνάδουν με τις υφιστάμενες διμερείς συνθήκες, τότε δεν θα υπάρξει επαρκής υποστήριξη για τις συμφωνίες της Ένωσης. Έτσι λοιπόν θα υπάρξει σημαντική καθυστέρηση της ε, πολιτικής της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν θα υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά των κρατών μελών ή των επενδυτών για να μεταβούν στο καθεστώς ε, των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ευρεία ισοδυναμία. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι οποιαδήποτε συμφωνία σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν μπορούν να ε, είναι πιο ακριβεί ε, σε ό,τι αφορά το καθορισμό του πεδίου τη προστασία των επενδυτών. Υπάρχει απόκληση απόψεων από αυτού, αλλά θα μπορούσε να πει κανεί ότι αν ε, δούμε την εξέλιξη των BITS, ε, οι χώρες που είχαν ε, πολλή εμπειρία με τις διαφορές προσπάθησαν να είναι πιο ακριβείς ως προς τον προσδιορισμό της προστασίας του επενδυτή. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι μιλάμε για μείωση του επίπεδου προστασίας, αλλά Απλά μιλάμε για ε, την αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογή των υφιστάμενων διατάξεων. Τώρα, αν επιτρέπει η συνθήκη της Λισαβόνα στην διατήρηση των υφιστάμενων beats. Ε, υπάρχει νομική συζήτηση από ό,τι φαίνεται από αυτού. Προσωπικά εγώ πιστεύω ότι η συνθήκη της ε, Λισαβόνας κάτι θα πρέπει να σημαίνει το ότι συμπεριλαμβάνεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να κινηθούμε πιο προ ολοκληρωμένες συμφωνίες και αυτό είναι και το όφελος. Αυτό είναι το όφελος, ε, ότι δηλαδή ενδυναμώνει τη θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση από την αποκλειστική αρμοδιότητα και υπάρχει και διευρυμένη πρόσβαση αλλά και επηρεάζει την εξέλιξη της επενδυτικής πολιτικής διεθνώς. Πιστεύω λοιπόν ότι η συνθήκη της Λισαβόνας ε, συνιστά μια αλλαγή και αντί να επικεντρωθούμε σε επιμέρους σημεία, ίσω θα πρέπει να δούμε καλύτερα τα ωφέλη που θα προκύψουν από τις συνολικές και καθολικές συμφωνίες, αν θέλετε. Η τρίτη σα ερώτηση είχε να κάνει με το πώς ε, μπορούμε να αποτρέψουμε τα κράτη-μέλη να μπλοκάρουν τη διαδικασία της μετάβασης. Και εδώ μπαίνουμε στην ουσία των ε, συμφωνιών ε, αυτών των μεταβατικών πρέπει να βρούμε έναν διακανονισμό, μια διευθέτηση που να, ασφαλίζει, να εξασφαλίζει η ασφαλεία δικαίου. Και πολύ σωστά αναφερθήκατε στο θέμα της παρεμπόδισης της εξέλιξης της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτό είναι το κύριο ζήτημα. Τι κριτήρια θα χρησιμοποιούσατε για την λήψη μια σχετικής απόφασης όταν ε, μία μπίτ κράτους μέλους ε, ε, καθορίζει την εξέλιξη της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν κάποιες διατάξεις πλατφόρμας, υπάρχει μια μπιτ κρατου μελους καθοριζει την εξελιξη της πολιτικη της ευρωπαικης ενωση υπαρχουν καποιες διαταξεις πλατφορμας υπαρχει μια συμπεφωνημενη πλατφορμα για τι επενδυτικέ πολιτικέ, αλλά δεν έχουμε ένα πανευρωπαϊκό μοντέλο για την BIT, ούτε υπάρχει τέτοια φιλοδοξία. Έτσι λοιπόν, αφόσον υπάρχει έλλειψη τέτοιου μοντέλου, πώς ε, προσδιορίζεται για το αν, το αν παρεμποδίζεται η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ίσως ε, αν υπάρξει εντολή διαπραγματευτική ε, για να διαπραγματευτείτε με ένα συγκεκριμένο εταίρο, θα μπορούσε αυτό να το χρησιμοποιήσετε ως κριτήριο. Γι' αυτό μια εναλλακτική θα ήταν να δεκτούμε ότι η διαδικασία είναι εν εξελίξη και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλα τα μέρη θα πρέπει να έχουν ένα ρόλο στο να διαμορφώσουν την εξέλιξη αυτή. Δηλαδή να επικεντρωθούμε στη διαδικασία και όχι να στοχεύσουμε στο να έχουμε ένα συγκεκριμένο μοντέλο για αυτές τις ε, διμερείς επενδυτικές συμφωνίες ε, και αναφερθήκατε και σε στόχους ε, αναπτυξιακούς αλλά και σε άλλους στόχους πολιτικές. Εγώ δεν αναφέρθηκα ιδιαίτερα στην εισαγωγή μου στα θέματα αυτά. Ένα από τα θέματα που μας απασχολούν εδώ είναι τον θα έπρεπε να υπάρχει ένα γενικό προήμιο σε οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να έχουμε διατάξει ουσιαστικού δικαίου. Έχουμε δει διατάξει ουσιαστικού δικαίου στις ε, συμφωνίες ελευθερών συναλλαγών τη ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσατε να σκεφτείτε ένα τέτοιο μοντέλο. Για τον κύριο Ρίφ, για το επίπεδο των λεπτομεριών. είναι κάπως δύσκολο το θέμα αυτό, γιατί πρέπει να κρίνει κανείς για το ποιο θα είναι ενδεχομένως ο μελλοντικό αντίκτυπος. Δηλαδή τι θα γίνει στο μέλλον, ε, θα αντιμετωπίσει περισσότερες ε, ε, υποθέσεις διαφορών η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί κάποιοι είπαν ότι δεν υπήρξαν πολλές τέτοιες περιπτώσεις μέχρι τώρα, δεν υπήρξαν πάρα πολλές προσφυγές κατά ε, κρατών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, έτσι λοιπόν αυτό τι σημαίνει ότι δεν είναι ευάλωτη σε αύξηση τέτοιων υποθέσεων. ή ναι, ε, δεν υπάρχει αύξηση των ροών. Ε, γιατί κοιτάξτε, εδώ αυτό πρέπει να το συνδέσουμε με την δυναμική στις αγορές. Έτσι λοιπόν η ερώτηση είναι πώς θα ε, αναπτυχθούν ε, οι μελλοντικέ επενδυτικές ροές στο μέλλον. Αν υπάρξουν μεγαλύτερες επενδυτικές ροές από τις άλλες χώρες μπορείτε να δείτε και άνοδο αυτών των διαφορών. Έτσι λοιπόν τότε ναι, μπορεί να χρειαστεί να μπείτε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Έχετε ένα σχετικό επιχείρημα. Το θέμα είναι πώς κρίνετε την εξέλιξη των διεθνών επενδυτικών ροών στις αγορέ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπερνασκόνη. Ευχαριστώ πολύ. Για το θέμα της διαφάνειας καταρχήν. Πιστεύω ότι η διαφάνεια <laughs> μπορεί να υπάρχει υπέρ όλων, δηλαδή και για τους πολίτες και για τους επενδυτές και για το κράτος υποδοχής των επενδύσεων για όλους. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος ε, του οποίους ε, θα δημοσιεύεται τις διαδικασίες ε, για διαφορετικό σκοπό. Από ό,τι φαίνεται, ε, όλα είναι σαφή. Σε διεθνείς υποθέσεις μπορείτε όλα να τα βρείτε online, επιγραμμικά. Και ξέρετε, όταν υπάρχουν ε, εμπιστευτικές πληροφορίες μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Δηλαδή αυτό το κάνουμε ήδη. Δεν υπάρχει λόγος, εφόσον το πράττουμε σε, εθνικό επίπεδο, να μην το κάνουμε και εδώ. Το όλο σύστημα προήρθε από ένα background εμπορική ε, επίλυσης διαφορών και δεν αρμόζει σε αυτό το μηχανισμό επίλυσης διαφορών. Τώρα, μπορούμε να δούμε τι έγινε με το chilling effect, αν υπάρχει τέτοιο αποτέλεσμα ή όχι, δεν το ξέρουμε. Πολλέ υποθέσει έχουν διευθετηθεί. Δείτε, παραδείγματο χάρη, τη συνεχιζόμενη υπόθεση κατά τη Γερμανία, όπου ένα Σουηδό επενδυτή, η Vattenfall, μείνησε τη Γερμανία για 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν ε, γνωρίζουμε εγώ δεν έχω καμία ιδέα τι συνέβη με την υπόθεση. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι υπάρχει γιατί κατατέθηκε υπό την EXIT, το οποίο έχει ένα σύστημα καταχώρησης και ξέρουμε ότι έχει ε, ανοίξει υπόθεση. Τώρα, αν καλύπτεται από ε, το δίκαιο του ΙΕΝ, ε, είναι υπό το διεθνές... Ε, ε επιμελητήριο από το επιμελητήριο της Στοκόλμης αυτό το είναι εντελώς μυστικό. Ε, έτσι λοιπόν, ε, τι έκαναν ο Καναδάς και είπα, έβαλαν στις συμφωνίες τους ότι όλα πρέπει να είναι διαφανή. Γι' αυτό γνωρίζουμε τι συνέβη στις υποθέσεις ναύτα. Και δεν είναι σωστό ότι υπήρξαν μόνο δύο περιπτώσεις. Σας έδωσα και το παράδειγμα με την Έθιλ. Είχαμε μια περιβαλλοντική υπόθεση εκεί και πλήρωσε ο Καναδάς και κατεργήσε και την νομοθεσία που νομοθεσία η οποία έμεινε ενισχύ σε άλλε χώρε όπω και στη ΣΥΠΑ. Τώρα, σε ό,τι αφορά λοιπόν αυτό το chill effect, είναι δύσκολο να έχουμε βάση δεδομένων. Μπορούμε να το ρυθμίσουμε στις συμφωνίες ε, και στην ΣΥΤΡΑΛ. Ε, ε, τώρα η Κομισιόν συμμετέχει στην Ασιτράλ, υπάρχει μια διαδικασία αναθεώρησης, ανεξελίξη, τα κράτη-μέλη, ε, πολλά κράτη-μέλη μπλοκάρουν τη διαφάνεια σε αυτή τη διαδικασία, όμως δεν ξέρω τι θα γίνει εκεί. Τώρα, αν υπάρχει όμως αναφορά στην on τράλ στις ε, συνθήκες και αυτοί οι κανόνες είναι πιο διαφανείς, τότε το όλο σύστημα θα καταστεί πιο διαφανές. Εγώ πιστεύω ότι αν για το μέλλον η πολιτική, αν θέλετε μια πολιτική διαφανές μπορείτε να συστήσετε ένα σύστημα και για ε, τα ένδικα μέσα. Δεν είναι εύκολο, αλλά θα μπορούσατε να το σχεδιάσετε. Τώρα σε ό,τι αφορά τις παλιές bit, ε, δεν νομίζω ότι θα συνεχίσουν να είναι μη διαφανείς, ακόμη και αν συνεχίσουν να ισχύουν ως προς την ουσία τους. Γιατί δεν θα έπρεπε το Κοινοβούλιο να γνωρίζει τι γίνεται στα κράτη-μέλη αν ε, η Ένωση έχει αρμοδιότητα για τα θέματα αυτά. Αυτά τα πράγματα πρέπει να καταστούν πιο διαφανή και πραγματικά απευθύνω έκκληση και είναι υπέρ όλων εκτός από των δικηγόρων που θέλουν να ε, διατηρούν για τον εαυτό τους πληροφορίες γιατί μπορούν να τις πουλήσουν πολύ ακριβά. Έτσι λοιπόν, εγώ θα υποστήριζα τη διαφάνεια. Σε ό,τι αφορά τώρα την ερώτηση για το πώς ε, αποφεύγουμε κοινωνικές και εμπορικές πολιτικές να προσβληθούν. Ε, συγγνώμη που θα πάρω το παράδειγμα τον είπα και πάλι. Ε, ξέρουμε ότι υπό την ΑΦΤΑ, μετά την ΑΦΤΑ κατατέθηκαν όλες αυτές ε, οι μηνύσεις ε, και τα μέρη έκαναν κάποιες ε, δηλώσεις ερμηνείας για να πούν τι εννοούν. Και μόνο πρόσφατα είχαμε ε, απόφαση επί μιας περιβαλλοντικής υπόθεσης ε, γκλάμις κατά Ηνωμένων Πολιτειών αφορούσε ένα ε, ανοιχτό ορυχείο και εκεί λάμβανε χώρα μια ε, μεγάλη επιχείρηση όταν ε, μήνυσε, μήνυσε ο επενδυτής ε, την Καλιφόρνια επειδή υπήρξε απέκτηση backfilling και μπορεί να υπήρχε δυνατότητα να χάσουν αν δεν είχαν κάνει αυτή την ερμηνεία τα κράτη, οι πολιτείε και έλεγαν ορίστε τι εννοούμε με το fair and equitable, με το δίκαιο, με τη δίκαιη μεταχείριση. Έτσι λοιπόν είναι θέμα ερμηνεία. Είναι σημαντική διατύπωση λοιπόν η γλώσσα που χρησιμοποιείτε. Αν θέλετε στο μέλλον να αποφύγετε να ε, να αποφύγετε τις διαδικασίες. Αν θέλετε να επηρεάσετε τις αποφάσεις, πρέπει να το δηλώσετε από πριν. Τώρα, για την περισσότερη μικρότερη προστασία, δεν νομίζω ότι μια όριστη ρήτρα σημαίνει ότι θα υπάρχει και μεγαλύτερη προστασία, γιατί δεν ξέρετε πώς θα αποφασίσει ο διαιτητής τελικά. Νομίζω ότι απάντησα τις ερωτήσεις και μακρηγόρησα και κάπως. Σας ευχαριστώ. Thank you for your Ευχαριστούμε για την εξαιρετική διαφάνεια. Ο καθηγητής Τίτιε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εφτά παρατηρήσεις θα αναφέρω. Πρώτον, για την ερώτηση για τα πρότυπα στο μέλλον της προστασίας, για τις απαλωτριώσεις και άλλα θέματα. Η απάντηση για μας, τους Ευρωπαίους, είναι απλή. Τα πρότυπα που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αν δούμε την ε, νομολογία των διαιτητικών δικαστηρίων για τις απαλωτριώσεις, βλέπουμε πόσο επηρεάζεται από την ομολογία του δικαστηρίου του Στρασβούργου. Είναι παρόμοια η προσέγγιση όπως ε, από το ε, δικαστήριο του Στρασβούργου με βάση το πρωτόκολλο 1 και σε μεγάλο βαθμό οι αποφάσεις των διαιτητικών δικαστηρίων ερμηνεύονται με τρόπο που συνάδει με την καλή διακυβέρνηση και τους κανόνες της ε, στο χάρτη ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης, επίσης, έτσι λοιπόν έχουμε ένα βασικό αν θέλετε υπόδειγμα που μας καθοδηγεί και έτσι διευκρινίζεται στην Ευρωπαϊκή Νομική Παράδοση του κράτους δικαίου. Δεύτερο ερώτημα αν με τη μεταφορά και μόνο της αρμοδιότητας, τα Μπιτς, που είναι διμερείς δηλαδή επενδυτικές συμφωνίες των κρατών μελών, καθίστανται ε, παράνομες. Θα ήθελα να τονίσω ότι όχι, δεν συμβαίνει αυτό, αυτή είναι η νομική μου άποψη. Μόνο και μόνο επειδή υπάρχει μεταβίβαση αρμοδιότητας, δεν επηρεάζει την νομιμότητα των BITS. Εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα είχαμε σοβαρά προβλήματα σε πολλούς τομείς, όπου τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ε, έμεσα ε, που οδήγησε σε ε, αποκλειστική αρμοδιότητα στο αστικό δίκαιο, στο οικογενειακό δίκαιο, στους ανοιχτούς ουρανούς όπου σιγά σιγά εμέσως απέκτησε αρμοδιότητα η Κομισιόν. Αυτό δεν επηρέασε συνθήκες και συμφωνίες των κρατών μελών. Επίσης, Μιλάμε για συγκεκριμένες διατάξεις που συγκρούονται, αλλά όχι, δεν, δεν θίγουμε την ομιμότητα των συμφωνιών αυτών, των BITS καθ' αυτών. Και θα πρέπει να δούμε τις δράσεις βάσει των συνθήκων. Επίσης, ένα δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τις, ε, για τις επενδύσεις σε αντιπαράθεση με τα διαιτητικά. Είναι ενδιαφέρουσα αυτή η προοπτική ενός διεθνούς ή περιφερειακού δικαστηρίου σε αντιπαράθεση με τα διαιτητικά δικαστηρία. Αλλά είναι, δεν είναι ρεαλιστικό. Από νομικής αυτό πρέπει να πούμε, διότι θα χρειαζόταν ήδη πολυμερή ε, συμφωνία, σε πολυμερή βάση, διεθνή συμφωνία ή σε περιφερειακή βάση. Υπάρχει το πρόβλημα της αμοιβαιότητας, γιατί για παράδειγμα να θέλει να μηνυθεί ο Καναδάς στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ποτέ δεν θα συμφωνούσε σε κάτι τέτοιο. Οπότε υπάρχει ένα προακτικό πρόβλημα που προκύπτει από τα νομικά αυτά θέματα και η καλύτερη προσέγγιση θα ήταν η μεγαλύτερη διαφάνεια και διαφάνεια στις διαιτητικές διαδικασίες και να δούμε και θέμα αυτά που αφορούν, αν θέλετε, την επιλογή των διαιτητών, δικαστών κλπ. Τώρα, το άλλο θέμα, γενικότερο αυτό, γιατί να επιτρέπετε σε μια επιχείρηση να μηνύσει μια κυβέρνηση, ένα κράτος. Και πάλι σας υπενθυμίζω τη νομική παράδοση εδώ. Εμείς εφεύραμε αυτό το θέμα, αυτή την ιδέα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι βασικό αυτό στο κράτος δικαίου στην Ευρώπη, ότι τα άτομα μπορούν να μηνύουν κυβερνήσει και δυνάμει της συνθήκη ε, σε σχέση με τα εμπορικά συμφέροντα αλλά και στα πλαίσια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οπότε νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρώπη γενικότερα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι μια πολύ καλή απάντηση στο ερώτημα γιατί μια επιχείρηση να μπορεί να μηνύσει την κυβέρνηση. Πέμπτο ερώτημα. Πρέπει να δεχτούμε όλες τις επενδύσεις όχι εδώ, δεν μιλάμε για πρόσβαση στην αγορά. Είμαστε ελεύθεροι να αποφασίζουμε ποιους θα δεχτούμε, ποιους ξένους επενδυτές θα δεχτούμε στην ε, εσωτερική και στην κοινή αγορά. Η ναύτα είναι ένα παράδειγμα. Βέβαια η γλώσσα ε, είναι σημαντική για ένα νομικό, από την άλλη όμως δεν ε, υπάρχει απόδειξη ότι οι μακροσκελέστερες διατάξεις συνεπάγονται μεγαλύτερη νομική ασφάλεια ως ένα βαθμό. Ε, παίζουν ρόλο διαφορετικές νομικές παραδόσεις ε, και ε, υπάρχει ευρωπαϊκή υπάρχει το αγγλοσαξονικό δίκαιο, η ευρωπαϊκή νομική παράδοση, η δικαιική παράδοση. Εδώ χρειάζεται προσοχή. Το έβδομο ερώτημα αφορά το αν ε, πρέπει να έχουμε ενιαία πρότυπα για τα bit των κρατών μελών. Αυτό θα γινόταν αν, υπήρξε, αν υπήρχε η ρήτρα πλέον ευνοουμένου κράτος, ε, κράτους. Ε, υπάρχουν κάποιες αποφάσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Ε, στηριζόμενοι στο διεθνές δίκαιο, δηλαδή τα κράτη-μέλη αφενός θα συνδέονταν μέσω κάποιας ε, συνθήκης ή παράγωγου δικαίου ε, σε σχέση με την, ε, το μάλλον ευνοούμενο κράτος που βέβαια θα προϋπέθεται και ε, συγκατάθεση του τρίτου κράτους σε βάση διεθνούς δικαίου. Αυτό αποτελεί ένα δύσκολο θέμα ε, σε διπλωματικό επίπεδο. Θα μπορούσε όμως να γίνει, όπως σας είπα, δυνάμει διεθνούς δικαίου. Και τέλος ο κύριος Adrian Van Den Hoffen. Πέντε λεπτά μάξιμου. Ευχαριστώ, θα κάνω ό,τι μπορώ κύριε Πρόεδρε να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις. Συμφωνώ με τον καθηγητή Τίτη εδώ, η συνθήκη της Λισαβόνας ε, δεν καθιστά παράνομα αυτομάτως τα μπίτσε Υπάρχουν όμως ρήτρες επιμέρους που γίνονται προβληματικές. Κάποιες από αυτές τις ρήτρες μπορεί να είναι πολύ σημαντικές. Οπότε ο κανονισμός κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια να δημιουργήσει νομική ασφάλεια γύρω από αυτές τις κεντρικής σημασίας ρήτρες για την προστασία των επενδυτών. Νομίζω όμως ότι μία από τις προκλήσεις αυτής της Επιτροπής βάσει του κανονισμού θα είναι να εξετάσει από κοντά μαζί με την Κομισιόν του εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, τους ειδικού για τις επενδύσεις, αυτό το σύστημα επανεξέτασης στο σχέδιο κανονισμού γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Το, η Business Europe δεν έχει όλες τις απαντήσεις, αλλά γνωρίζουμε τις ανησυχίες των κρατών μελών όταν καλύπτεται πολύ καλά από BITS, από σε εμερητικές συμφωνίες. Άλλες, μικρότερες χώρες δεν ωφελούνται γιατί δεν θα έχουν τέτοια κάλυψη μέσα από τα BIT. Από την άλλη πλευρά όμως, ε, ρισκάρουν οι επενδυτές αν ανασταλούν οι συμφωνίες. Τι θα γίνει λοιπόν στη συνθήκη της Λισαβόνα, υπάρχει υποχρέωση των κρατών μελών να συνεργάζονται. Ίσως αυτό θα μπορούσε να είναι ένα στοιχείο προβληματισμού, ένα πρίσμα μέσα από το οποίο θα το δει η Επιτροπή το θέμα και μαζί με τα κράτη-μέλη θα ε, λύσει αυτά τα μεγάλα προβλήματα. Τώρα, για το policy space, ε, πολιτικός χώρος για τις κυβερνήσεις, το ρυθμιστικό πάγωμα, το regulatory chill που αναφέρθηκε και το έθεσε και, και η κυρία Μπερνασκόνη. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην ε, είμαστε υπερβολικά αμυντικοί. Υπάρχει ε, ο προβληματισμός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα περιοριστεί στην δυνατότητά της να υιοθετεί κοινωνική νομοθεσία, περιβαλλοντική νομοθεσία ή οποιαδήποτε νομοθεσία. Αλλά η εμπειρία μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει ότι ούτε ο ΠΟΕ Ούτε οι διμερείς επενδυτικές συμφωνίες, τα BITS ή άλλες διεθνείς συμφωνίες δεν περιόρισαν την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τώρα. Έχουμε προχωρήσει σε όλα αυτά τα μέτωπα και στο περιβάλλον και σε ένα σωρό άλλους τομείς. Εκεί που υπάρχει περιορισμός είναι ότι δεν επιτρέπεται να κάνουμε διακρίσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξένους Ευρωπαίους και ξένους επενδυτές. Αυτός είναι ένας πολύ σοβαρός και αυστηρός περιορισμός, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε διακρίσεις. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να αντιταχθούμε στην αρχή αυτή που είναι μια βασική αρχή ε, και η οποία συνάδει με το κράτος δικαίου στην Ευρώπη. Από την άλλη πλευρά έχουμε εμπειρία και τα μέλη της Επιτροπής αυτής γνωρίζουν πολύ καλά ότι ορισμένοι εμπορικοί μας εταίροι εφαρμόζουν με διακριτικό τρόπο το δικό τους δίκαιο. Είχαμε πρόσφατα προβλήματα με την Κίνα σε σχέση με την εφαρμογή του δικαίου για την πνευματική ιδιοκτησία, ε, την νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις, τα προβλήματα με τη Ρωσία και το περιβαλλοντικό δίκαιο που εφάρμοσε με διακριτικό τρόπο σε βάρος των επιχειρήσεων εταιριών μας. Αυτή είναι η εξαγωγική πλευρά των επενδύσεων και η προκλήση που αντιμετωπίζουμε. Γι' αυτό χρειαζόμαστε την προστασία των BITS, των διμερών επενδυτικών συμφωνιών και των επενδυτικών συμφωνιών της ευρωπαϊκή Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει λοιπόν να είναι πιο εξωστρεφής, όχι εσωστρεφής. Ένας άλλος λόγος για τους οποίους δεν έχουμε προβλήματα σε βάρος Ευρώπη, Ευρώπης είναι γιατί σπάνια οι ευρωπαϊκές ε, χώρες κάνουν απαλωτριώσεις και όταν κάνουν για να περάσει ο σιδηρόδρομος, μια γραμμή ή κάτι τέτοιο, τότε υπάρχει, προβλέπεται καλή αποζημίωση. Ε, οι περισσότερες ε, επενδύσεις, ε, στις επενδύσεις πολλές φορές υπάρχουν προβλήματα όταν οι απαλωτριώσεις δεν προβλέπουν αποζημίωση. Για το θέμα της διαφάνειας και αυτό είναι ένα θέμα υποσυζήτηση από τη δική μας την πλευρά μπορούμε να δεχτούμε βελτίωση της διαφάνειας με την προϋπόθεση ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες θα προστατεύονται και με την προϋπόθεση ότι μόνο τα πραγματικά, τα γνησίως ενδιαφερόμενα μέρη, οι αμίκους κιούρε για παράδειγμα, θα μπορούσαν να συμμετέχουν σε τέτοιες διαιτησίες, γιατί δυστυχώς σε χώρες όπου δεν έχουμε την ελευθερία του συνεταιρίζεσθε, ελευθερία μη κυβερνητικών οργανώσεων. Έχουμε κυβερνητικές ε, οργανώσεις που είναι μη κυβερνητικές και παίζουν συγκεκριμένο ρόλο και εκεί θα ρισκάρουν, θα ε, εκτεθούν σε προβλήματα. Φαντάζεστε σε ποιες χώρες. Αυτά είναι κάποια από τα προβλήματα Αυτά από την πλευρά μου. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι θα πρέπει να ακούσουμε και τις αντιδράσεις των άλλων θεσμικών οργάνων, γιατί οι ακροάσεις ε, τους ενδιαφέρουν και τους άλλους. Οπότε ας δούμε ε, το Συμβούλιο που είναι παρόν. Παρακαλώ ένα σύντομο σχόλιο αν θέλετε. Ε, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε θα ήθελα, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, θα ήθελα να αντιδράσω στην παρέμβαση του κυρίου Στέντερ πριν από λίγο που έχει σχέση με τον ε, κανονισμό μετάβασης. Ε, μίλησε για την συνθήκη της Λισαβόνας η οποία δεν επιτρέπει το status quo αλλά φοβόταν το μποϊκοτάρισμα από πλευράς κρατών μελών και είπε ότι ε, θα πρέπει να υπάρξουν διμερείς συνθήκες οι οποίες ή να επανασυζητηθούν ή να αποσυρθούν τελείως. Το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι ότι πρέπει να είμαστε απόλυτα ρεαλιστές σε, την, αυτό το θέμα γιατί εάν υπήρχε μια λύση η οποία από τη μια μέρα στην άλλη ε, μας επέτρεπε να αντικαταστήσουμε όλα αυτά τα παράβλευρα τα οποία έχουν και διάφορες διατάξεις θα υπήρχε πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι στην πράξη η επαναδιαπραγμάτευση των συμφωνιών είναι χρονοβόρα και ε, είναι κάτι πολύ σημαντικό που είπαμε επίσης εδώ είναι και το τρίτο μέρος. Το τρίτο μέρος θα θέλει την επαναδιαπραγμάτευση για να αλλάξει ένα σημείο μέσα στην συμφωνία. Αυτό το βλέπουμε και σε άλλους τομείς. Ε, Παραδείγματο χάρη μεγάλοι γείτονες, μεγάλοι εταίροι για μια ε, συμφωνία εταιρικότητας την οποία θέλουμε να επαναδιαπραγματευτούμε για το θέμα της ενέργειας. Ένα θέμα πολύ ευαίσθητο για μας. Ε, δεν τα καταφέρνουμε λοιπόν να, να ανανεώσουμε αυτή τη συμφωνία γιατί εμάς μας ενδιαφέρουν οι επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα που είναι πολύ ευαίσθητος αυτό υπόθηκε και πριν από λίγο οπότε όπως υπογραμμίσαμε ε, ε, ε, ισχύουν οπωσδήποτε συνεχίζουν να ενισχύουν οι διεθνείς συμφωνίες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο εφόσον υπάρχει δέσμευση στην συνθήκη της Λισαβόνας υπάρχει και προσανατολισμός στο μέλλον το καλύτερο θα ήταν ε, βεβαίως να υπήρχε επαναδιαπραγμάτευση. Αυτό θέλουμε. Αλλά αν οι διμερείς συμφωνίες καμιά φορά δίκαια λέμε, επειδή έχουν παλιώσει, επειδή προέρχονται από άλλο τομέα, δεν είναι προσαρμοσμένοι λοιπόν στις πολιτικές ε, απόψεις της στιγμής, παρόλο που δεν είναι τέλεια, υπάρχει όμως μία προστασία, προστασία νομική. Οπότε ας μην τις απειλήσουμε αυτές τις ε, συμφωνίες γιατί δεν έχουμε λύσεις έτοιμες για να τις αντικαταστήσουμε μια ανοιχτή. Οι ανησυχίες του, των κρατών μελών είναι οι εξής. Έχουμε νομική ασφάλεια, υπάρχουσα, ε, όμως ε, με πολύ θεμητές ιδέες υπάρχει αυτή η ασφάλεια που θέλουμε να δώσουμε είναι νέα, αλλά θα πάρει πολύ χρόνο η αλλαγή της. Παραδείγματος χάρη οι διμερείς συμφωνίες παίρνουν χρόνια. Εάν δούμε για ένα κράτος μέλος που μετά από 9 χρόνια με ένα μεγάλο εμπορικό εταίρο, μια αφρικανική χώρα, θέλησε να συνάψει μια συμφωνία διμερή και πήρε 9 χρόνια η όλη διαδικασία. Λοιπόν, ας είμαστε πραγματιστές, να το ξέρουμε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την ε, Προεδρία του Συμβουλίου της Ένωσης. Ε, επίσης θα ήθελα να ακούσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια τελική σύντομη παρατήρηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα πράγμα θέλω να πω για το θέμα της ισχύως των ε, λεγόμενων των τριών ε, ομιλητών. Είναι δύσκολο να πούμε γιατί το πράττουμε αυτό. Κανείς δεν διαφωνεί με τις, ε, την ισχύουσα αξία αυτών των συνθήκων που ισχύουν σύμφωνα με το υπάρχον δίκαιο. Το θέμα είναι τι υποχρεώσεις έχουν τα κράτη-μέλη μετά από τη Λισαβόνα. Εδώ υπάρχει αβεβαιότητα και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα πίστευε ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε να επικρατήσει αυτή η αβεβαιότητα. Αυτό είναι ένα ξεχωριστό θέμα πέρα από το περιεχόμενο των συνθήκων. Ο προταθής κανονισμός δεν γιατρεύει τα σημεία όπου υπάρχει ασύμβατος χαρακτήρας με τις συνθήκες το να υπάρχουν και να συνεχίζουν να υπάρχουν οι κανονικές διαδικασίες και να εφαρμόζονται, ναι, αυτό το έχει χαιρετήσει σε ορισμένες περιπτώσεις όταν ήταν απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ας μην επικρατεί όμως σύγχυση. Άλλο η ισχύ αυτών των ε, συμφωνιών σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και άλλο είναι η μεταβατική περίοδος πάρα πολύ συγκεχημένη, πάρα πολύ σύνθετη και η οποιαδήποτε αλλαγή στην κατάσταση την οποία θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να την επιλύσει ως πρόβλημα με τον ΑΒ τρόπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εγώ τους φιλοξενουμένους μας ε, οι οποίοι μας έδωσαν μια πληρέστατη εικόνα, μια θετικότατη συμβολή. Στο, φτάσαμε στο πέρας αυτής της ακρόασης στο, και είμαστε πολύ καλύτερα πληροφορημένοι τώρα από ό,τι ήμασταν προηγουμένως σχετικά με τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και οι οποίες βρίσκονται μπροστά στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ και πάλι. Θα περάσουμε τώρα στο θέμα 16 ας ε, περάσουν έξω όσοι θέλουν να βγουν. The so that you can... Παρακαλώ, παρακαλώ βοηθήστε μας να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να ανακαινώσετε την αίθουσα χωρίς θόρυβο στο μέτρο του δυνατού παρακαλώ πάρα πολύ ήσυχα και γρήγορα. And also may not και σας παρακαλώ μην συζητάτε στο ιστορικό της αίθουσας. Please, may I have attention, please. We need to go on. We have just one hour for the next four items. Έχουμε μία στη μας για τα επόμενα τέσσερα σημεία. Δεν ε, είμαι σίγουρος ότι προλαβαίνουμε να τα εξετάσουμε, αλλά ας προσπαθήσουμε. Ας ξεκινήσουμε με το σημείο 16. Η μηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης. Εδώ έχουμε ένα σχέδιο γνωμοδότησης ε, από τον Τζαν Λούκα Σούστα, από τους σοσιαλιστές. Και θα συζητήσουμε τώρα το σχέδιο γνωμοδότησης. Η ε, η μηχανική πολιτική και η εμπορική πολιτική θα πρέπει να αλληλοποστηρίζουν η μία την άλλη και μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης είναι μία από τις θεματικές πρωτοβουλίες ε, υπό τη στρατηγική της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020. Τώρα, πώς μπορεί η εμπορική πολιτική να βοηθήσει την Ευρώπη να επωφεληθεί για την ε, ε, ανάπτυξη της οικονομίας και πώς μπορούμε να έχουμε μια βιομηχανική πολιτική στην εποχή της πυγκοσμοποίησης. Αυτά είναι τα θέματα που καλούμαστε να συζητήσουμε. Τζαν Λούκα, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ. Give me Please do not hold conversations in the... παρακαλώ, αν θέλετε να συζητήσετε, παρακαλώ εκτός της αίθουσας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα, γιατί δεν έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας και γιατί είχαμε ούτως ή άλλως μια καλή ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μας πριν λίγες εβδομάδες. Αυτή η ε, έκθεση απευθύνεται και στην Επιτροπή Ήτρε, που είναι και μέλος αυτής της Επιτροπής ε, και προέρχεται και από τη δική μου ομάδα. Εδώ αναφερόμαστε στην βιομηχανική πολιτική στο πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου. Έτσι λοιπόν, στον δυνατότητα που έχουμε να αναλάβουμε δράση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προσπαθήσαμε να δούμε ποιες είναι, ποιοι είναι οι κυρίοι στόχοι και έτσι λοιπόν έχουμε τονίσει τη σημασία της βιομηχανικής πολιτικής λαμβάνοντα υπόψη ότι τουλάχιστον ε, τα τελευταία 15-20 χρόνια εμεί είδαμε μια προοδευτική ενίσχυση των υπηρεσιών εις βάρος του βιομηχανικού τομέα, του δευτερογενούς δηλαδή και του πρωτογενούς τομέα, του αγροτικού τομέα, αλλά ο τομέας των χρηματο-οικονομικών και χρηματοπιστωτικών περισσιών ε, δεν θα πρέπει να ακυρώσει ένα σημαντικό πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής εμπορικής πολιτικής, δηλαδή της βιομηχανίας και αναφέρομαι κυρίως στην μεταβητική βιομηχανία ποιότητας, ε, η οποία προσανατολίζεται προς την εφορία και αντιμετωπίζει και τις περιβαλλοντικές προκλήσεις που μας παρουσιάζονται σε αυτόν τον κόσμο και έχει ως στόχο να διατηρήσει και τις θέσεις εργασίας, ιδίως μετά την ε, χρηματοπιστωτική κρίση. Μπαίνει ε, λοιπόν εδώ και το θέμα της ε, οικονομικής εξυγίανσης και της μείωσης του χρέους. Ε, μπορώ να σας πω ότι είναι σημαντικά αυτά τα θέματα για να μπορέσει να παραμείνει η πιο μεγάλη οικονομία του κόσμου, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο πιο μεγάλος οικονομικός χώρος στον κόσμο. Έτσι λοιπόν ζητάμε στην έκθεση ε, να υπάρξει υπεράσπιση των πνευματικών δικαιωμάτων, ενίσχυση των περισσοκών στοιχείων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, να απελευθερωθούν οι προστατευμένες αγορές. Συζητήσαμε εδώ και δύο ώρες για τις επενδύσεις στις παγκόσμιες αγορές, για τη σταθεροποίηση των συναλλαγών και το ότι σήμερα βλέπουμε μια πολιτική συναλλαγών η οποία δεν είναι στο ύψος αυτής της παγκόσμιας αγοράς που εμείς επικαλούμαστε. Ας ε, δούμε τι γίνεται και στις συναλλαγές με την Κίνα. Επίσης αναφερόμαστε στην ε, νομική προστασία των επιχειρήσεων στο εσωτερικό, στην καταπολέμηση της παραποίησης ε, και στην καταπολέμηση του αθεμίτου του ανταγωνισμού. Έτσι λοιπόν η βιομηχανική πολιτική χρειάζεται αυτό το πλαίσιο κανόνων και υποστήριξης και η χρηματοοικονομικής υποστήριξης, γιατί το δικό μας βιομηχανικό και παραγωγικό σύστημα πρέπει να μπορεί να είναι ανταγωνιστικό στις παγκοσμίες αγορές. Θα παρουσιαστούν και τροπολογίες επιτυχίε τις επόμενες ημέρες και ελπίζω να μπορέσουν να μα βοηθήσουν στο να βελτιώσουμε αυτή τη βάση συζήτησης ε, που οικοδομείται βάσει της έκθεσης. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση του σχεδίου γνωμοδότησης. Έχετε το κείμενο στο φάκελό σας. Όπως μας επενθύμησε και ο συγητής, πρόκειται για μια συνεισφορά στο φάκελο Ήτρε. δηλαδή στην ε, αρμόδια Επιτροπή Βιομηχανίας αυτού του Κοινοβουλίου. Να δώσω το λόγο σε άλλα μέλη της Επιτροπής μας που μπορεί να θέλουν να κάνουν κάποια σχόλια. Όχι, ας περάσουμε στην Κομισιόν. Ο κύριος Μπέρκμαν από τη Διεύθυνση Βιομηχανίας. Ευχαριστώ πολύ. Καλωσορίζουμε το σχέδιο έκθεσης από τον κύριο Λάγκε Φαίνεται ουσιαστικά να είμαστε στο ίδιο μήκο κύματο εδώ. Αν μου επιτρέπετε, χρειάζεται η Ευρώπη μια ισχυρή και ανταγωνιστική βιομηχανική βάση. Οι μεταποιητές μας πρέπει να, πρέπει να ε, δρούν ε, βάσει δύο κανόνων με τους διεθνείς ανταγωνιτές τους. Επίσης εκτιμούμε το ότι συζητείται αυτό το θέμα και σε αυτήν την Επιτροπή και ότι αυτή η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι βιομηχανική πολιτική ως ζωτική σημασία για την ε, εμπορική πολιτική. Επίσης θεωρούμε πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε τον ε, έντονο ανταγωνισμό από τους παγκοσμίους εταίρους μας και πρέπει να ενδυναμώσουμε την Ευρώπη, πρέπει να βασιστούμε στο δύναμη που έχει, ότι έχει 20 εκατομμύρια επιχειρήσεις, 500 ε, εκατομμύρια κατοίκους ε, και πάρα πολλές ε, πάρα πολλά εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να εκτεθούμε στον αθέμητο ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα πρέπει να δούμε ε, ότι υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα στον κόσμο. Το δικό μας μοντέλο βασίζεται στο άνοιγμα των αγορών και σε κοινωνικές οικονομίες αγοράς, αλλά άλλα μοντέλα ανάπτυξη σήμερα ακολουθούν διαφορετικές προσεγγίσεις που σε κάποιο βαθμό επίσης συμπεριλαμβάνουν στοιχεία προστατευτισμού δηλαδή σε ό,τι αφορά την πρόσβαση των επενδύσεων στις αγορές, πρόσβαση στις αγορές για πώληση των αγωθών ή πρόσβαση των αγορών ε, πρώτων υλών. Και εκτιμούμε πάρα πολύ το ότι αυτή η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το λαμβάνουν αυτό δεόντως υπόψη και προσπαθούν να αναλάβουν εκ των προτέρων δράσεις για τη δημιουργία αυτού του καθεστώτος ε, ίσων κανόνων. Ανυπομονούμε να λάβουμε την έκθεση του Κοινοβουλίου και χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε συγκλίνουσες απόψεις από αυτού. Η Κομισιόν στις 28 Οκτωβρίου δημοσίευσε ένα έγγραφο για τη βιομηχανική πολιτική, από ό,τι καταλαβαίνω και το Συμβούλιο προσπαθεί να εξάγει συμπεράσματα για την πρόταση της Κομισιόν. Έτσι λοιπόν αναμένουμε και την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις αρχές του επόμενου έτου. Σας ευχαριστώ. Ναι, είναι οι ίδιες οι βασικές θέσεις των θεσμικών οργάνων. Ο κύριος... Α, δεν έχουμε άλλους. Η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι 11 του μήνα. Προχωρούμε. Σημείο 17. Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωργία και Διεθνές Εμπόριο. Η Επιτροπή Γεωργίας κάνει έκθεση δεύτερο πρωτοβουλία εμείς γνωμοδοτούμε για να συμβάλλουμε με βάση τη διαδικασία ε, των επιτροπών. Η συντάκτρια της γνωμοδότησης ε, από το ΕΛΚ, η κυρία Γκοντελιέβρο Κουίστχου Τρόβολ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Έχετε το σχέδιο έκθεσης όλοι, υπάρχει σε όλες τις γλώσσες. Οπότε μιλάμε επί τη βάση κειμένου πλέον. Πριν από την έκθεση αυτή προηγήθηκε συζήτηση με τον ε, εισηγητή από την Επιτροπή Γεωργίας και συνεννοηθήκαμε να επικεντρωθούμε ε, ο καθένας σε συγκεκριμένα θέματα, γιατί είναι μεγάλη θεματική γεωργία και διεθνές εμπόριο. Εδώ και δεκαετίες έχουμε το πρόβλημα ότι όταν βλέπουμε τη γεωργία μέσα από την εμπορική πολιτική, ταυτόχρονα υπησέρχονται και άλλα θέματα, συνειδητά ή όχι, όπως μικρή, ντόπιοι παραγωγή, αναπτυσσόμενες χώρες, χώρες ΑΚΕ, όλες οι χώρες με τις οποίες έχουμε προτιμησιακό σύστημα κλπ. Δεύτερον, στην νέα μας πολιτική των διμερών συμφωνιών, δηλαδή θέλουμε την τόχα, αλλά αφού δεν τα καταφέρνουμε πάμε από άλλο δρόμο, σε όλες αυτές τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών έχουμε συνιστώσεις γεωργικής πολιτικής. Αυτές οι συνιστώσεις είναι εντελώ ασυντόνιστες. Μιλάμε ξαφνικά με το Μερκοζούρ για τη ζάχαρη, για την μπανάνα με άλλους. Η δεξιά δεν ξέρει τι πει η αριστερά ο καθένας, ε, η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου λέει το Α, η ε, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας λένε το Β και θίγονται και οι γεωργοί μας και οι Πεθρός, που ούτως ή άλλως έχουν πολλά προβλήματα. Άρα, πρώτον, οριοθέτηση αρμοδιοτήτων των διαφόρων επιτροπών. Δεύτερο σημείο, πώς συνδυάζονται σε μας ε, η γεωργία και το εμπόριο. Εγώ έχω καταγράψει κάποια θέματα αρκετά γενικά, θα τα διαβάσετε μόνοι σας, γιατί δεν θα τα επαναλάβω εγώ εδώ. Επίσης, ε, δεν ε, παραθέτω παραδείγματα με μία εξαίρεση μόνο. Σκέφτηκα ότι όταν αρχίζουμε να παραθέτουμε παραδείγματα ε, ε, δεν καταλήγουμε πουθενά γιατί όλοι μας έχουμε εμπειρίες, όλοι μας στις διάφορες περιφέρειες έχουμε προϊόντα σημαντικά για μας. Η μόνη εξαίρεση είναι στο σημείο 3. Χαιρετίζει τη συμφωνία για το εμπόριο μπανάνας που διευθετεί διαφορές 20 ετών με τον ΠΟΕ. Πάντοτε σκεφτόμουν ότι αυτή η συμφωνία είναι εντάξει. Σήμερα το μεσημέρι συμμετέσχον σε μια ενημερωτική εκδήλωση για τις μπανάνες και την ε, οργάνωση της αγοράς για τις μπανάνες. Και η παραγωγή, που εγώ δεν τους ήξερα μέχρι τώρα προσωπικά, δεν φαίνονται ευχαριστημένοι. Έκπληξη. Μία ώρα αργότερα Ήρθαν οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας Ζάχαρης στο γραφείο μου και μίλησαν για τις συμφωνίες και τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με την Νότια Αμερική. Είχαν και αυτοί τις απαιτήσει τους. Το σημείο 3 για τις μπανάνες θα το κόψω λιγάκι και θα προσθέσω κάτι για τη ζάχαρη που είναι το προϊόν που επηρεάζεται πολύ από το εμπόριο. Κατά τα άλλα, σε όλη την έκθεση, καθ' όλη τη διάρκεια της ε, εργασίας μου, συνομιλούσα και με τους συναδέλφους από την Επιτροπή Γεωργίας, ε, ούτω ώστε να κινηθούμε παράλληλα λίγος πολύ και θα χαιρόμουν και εδώ στην Επιτροπή μας να δηλώσουν οι συνάδελφοι ότι είναι ικανοποιημένοι, αυτό θα ήταν ο ύψιστος έπαινος για μένα. Αν δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένοι, ας καταθέσουν τροπολογίες για να επιδιώξουμε συμβιβαστικές λύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τι λέγουν τα άλλα μέλη της Επιτροπής. Ο Τζιαν Λούκα από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες να σας πω και εδώ είναι τα άγχη ότι εγώ συμμερίζομαι με την άποψη της προλαλήσεως σας συναδέλφου. Συμφωνώ γιατί εδώ συμπεριλαμβάνω τα αρχές που αποτελούν ε, τη βάση της προσέγγισης που είχε πάντοτε η Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα της γεωργίας και της συνεισφοράς στο εμπόριο. Τώρα, τέσσερις διευκρινήσεις Καταρχήν, επί της ε, συμφωνίας για την μπανάνα, εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να δίνουμε κάπως μικρότερη έμφαση στο κείμενο. Δηλαδή, εντάξει, σημειώνουμε ότι είναι χρήσιμη αυτή η συμφωνία, αλλά τώρα να υπερβάλλουμε και να το παρουσιάζουμε πιο θετικό από ότι είναι, εγώ δεν θα το έκανα. Εγώ απλώς θα σημείωνα ότι υπάρχει μια συμφωνία που επιλύει ένα θέμα πολύπλοκο, αλλά θα έδινα μικρότερη έμφαση. Θα κάνω μια τροπολογία προς αυτήν την κατεύθυνση. Επίσης, έχουμε το θέμα ε, των πολυμερών και των διμερών σχέσεων. Νομίζω ότι και εδώ είναι μια κατάλληλη στιγμή για να επιβεβαιώσουμε εκ νέου ότι προτιμούμε τις ε, πολυμερείς σχέσεις ε, έναντι των διμερών, δυνάμει και των δυσκολιών που υπάρχουν στην Τόχα. Εγώ θεωρώ ότι και εδώ υπερβολικά δίνουμε έμφαση στη σημασία των διμερών συμφωνίων, ενώ το πρόβλημα της Γεωργίας αυτή τη στιγμή έχει σταματήσει γιατί στην Τόχα το βάρος της Γεωργίας και συγκεκριμένα του προστατευτισμού ε, από την Αμερικανική πλευρά μπλοκάρει τη συνέχιση των συζητήσεων του γύρου της Τόχα. Τρίτο στοιχείο, το θέμα της αμοιβαιότητας. Ε, αυτό υπογραμμίζεται, αλλά και αυτό ε, εδώ. ότι πάντως θεωρώ ότι με βρίσκει σύμφωνο το θέμα της αμοιβαιότητας που έχει να κάνει με την ποιότητα των προϊόντων, με τα πρότυπα, με την υγεία. Όλα αυτά ευνοούν ε, μεγαλύτερες συναλλαγές και με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ας ακούσουμε, Ας ακούσουμε τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. <clears throat> Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και την Επιτροπή σας για τις ε, προτάσεις αυτή την ε, γνωμοδότηση ε, σε σχέση υπάρχουν με, την έκθεση Παπαστάνκου ορισμένες ε, ε, σκέψεις οι οποίες υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σήμερα σημειώνουμε όλες τις προτάσεις που υποβάλλει και η δική σας Επιτροπή ούτως ώστε να δούμε για το πώς θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει τις ε, ε, διεθνείς ε, προδιαγραφές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν τώρα οι απαιτήσει της ΕΕ για τα διάφορα γεωργικά προϊόντα τα οποία θα τοποθετηθούν στην αγορά της ΕΕ και τα οποία θα πρέπει να συμμορφώνονται με την νομοθεσία της ΕΕ. Όλα αυτά αφορούν την ασφάλεια των ε, προϊόντων, την ευζοία και την υγεία των ζώων και σε σύμφωνη γνώμη με τις ε, προδιαγραφές της ε, υγιεινής ε, και της ασφάλειας, κάτι που δεν μπορούμε όμως να επιβάλλουμε στις τρίτες χώρες και δεν αντικατοπτρίζεται στις, στην ποιότητα των προϊόντων. Ε, παραδείγματος χάρη τα, οι προδιαγραφές που αφορούν την ευζοία των ζώων που δεν έχουν γίνει αντικείμενο ομοιομορφοποίησης από τον ΠΟΕ. Έχουμε λοιπόν συζητήσεις ανάλογες σε διάφορα φόρα διεθνή αντιστοίχως. ακολουθούμε τις ε, ε, διάφορες θέσεις του εισηγητή σήμερα για το πόσο ευαίσθητο είναι το θέμα της ζάχαρης σαν προϊόν σε όλες τις διεθνείς διαπραγματεύσεις και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να τα διατυπώσω αυτά κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ θέλει κανείς να υποβάλει τις τελικές παρατηρήσεις. Ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις συνάδελφε Σούστα. Δεν θα πρέπει να διαλέξουμε μεταξύ διμερών και πολυμερών ή να πούμε το ένα είναι καλό και το άλλο όχι, αλλά αντικειμενικά πρέπει να διαπιστώσουμε ότι οι διμερείς συμφωνίες δεν έχουν την ίδια συνέπεια, ιδιαίτερα εις ό,τι αφορά τα γεωργικά προϊόντα όπως ε, γίνεται με τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις και όταν περάσουμε από τις ε, πολυμερείς στις διμερείς, οι διμερείς θα πρέπει ξαφνικά να ισχύουν για όλους και αυτό δεν μπορεί να είναι προς το συμφέρον της γεωργίας. Ένα είναι αυτό. Αν όμως πιστεύετε ότι δεν είναι ισορροπημένο το κείμενο, με τα χαράς να το συζητήσουμε μαζί και να καταλήξουμε σε μια διαφορετική διατύπωση. Και καλό είναι να συμφωνήσει και η Κομισιόν. Για το σημείο 7, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν έχει δίκιο. Μπορούμε να ζητήσουμε πρότυπα, αλλά όχι να απαιτήσουμε και συγκεκριμένη διαδικασία. Αν όμως δεν ζητάμε συνεχώς βελτιώσεις, ιδιαίτερα από την προστασία των ζώων, της εργασίας του περιβάλλοντος, ε, από τα κράτη εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα αποδυναμώσουμε την δική μας ανταγωνιστικότητα, γιατί πρέπει να ανταγωνιζόμαστε κράτη με πολύ χαμηλούς μισθούς και ημερομίσθια. Πώς θα τις ανταγωνιστούμε. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε τα περιβαλλοντικά, τα κοινωνικά πρότυπα να έχουν διεθνή ισχύ. Σιγά σιγά, βήμα το βήμα, δεν μπορεί αυτό να είναι απόλυτη αξίωση, το καταλαβαίνω. και θα προσπαθήσω να βελτιώσω τη διατύπωση ε, στο σημείο αυτό. Ευχαριστώ. Η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι η 11 του μηνός. Σε λίγες μέρες δηλαδή. Ευχαριστούμε πολύ. Προχωρούμε στο σημείο 18 αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις έκτακτης ανάγκης για το Πακιστάν. Την περασμένη φορά ακούσαμε μία παρουσίαση του φακέλου αυτού από την Κομισιόν. Πολύ συγκεκριμένη είναι η φύση του πακέτου γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσημα επιδιώκει να αξιοποιήσει το εμπόριο ως εργαλείο. Την περασμένη φορά κάναμε κάποιες ερωτήσεις και μας απάντησε η Κομισιόν σε σχέση με το σκεπτικό της χρήσης του εμπορίου ως εργαλείου βοήθειας και αν αυτό αποτελεί προηγούμενο σε επόμενες ομιγέννητο φυσικές καταστροφές. Επίσης θα διαθέσει η Κομισιόν στην Επιτροπή της αξιολογήσεις που οπωσδήποτε θα έκανε σχετικά με τον αντίκτυπο των προτινομένων προτιμήσεων για το Πακιστάν. Επίσης υπάρχουν καθόλου ρήτρες διασφάλισης μετά τα προηγούμενα που είχαμε με άλλες περιπτώσεις μονομερών προτιμήσεων που χορηγήθηκαν για την αναδιάρθρωση, ανασυγκρότηση κάποιων χωρών. Και μπορεί να μας δώσει διασφάλιση κομισιών ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα στη Γενέβη με το ΓΚΑΤ και τις παρεκκλήσεις. Έχουμε ορίσει εισηγητή. Από την ελεύθερη συμμαχία, Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία. Και θα του δώσουμε το λόγο για να μας μιλήσει για τις βασικές γραμμές της μελλοντική έκθεσης του. Θα είμαι συντομότατος, όχι επειδή είναι το τέλος της μέρας, αλλά επειδή θέλω να ακούσω τους άλλους κυρίως. Είναι προφανές μετά από ένα χρόνο που είμαι εδώ. Η γνώμη μου και η γνώμη του κόμματός μου διαφέρει άρδιν επί πολλών θεμάτων από τα άλλα κόμματα και ομάδες. Σε αυτό το θέμα όμως επιζητώ τη μέγιστη δυνατή συμφωνία συνένεση να πω και προσβλέπω ίσως τη μέγιστη υποστήριξη από τα μέλη της Επιτροπής. Τα επιχειρήματα είναι σε δύο επίπεδα. Πρώτον, στο Πακιστάν είναι πολύ σοβαρή η ανθρωπιστική καταστροφή λόγω της πλημμύρας και της κλίμακας που προσέλαβε είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε το πρόβλημα. Πάνω από 2 εκατομμύρια εκτάρια καλλιεργιών καταστράφηκαν ή έπαθαν ζημιά και πάνω από ένα ε, και πολλοί αγρότες ε, χάθηκαν. 20 εκατομμύρια επηρεάστηκαν, 10.000 σχολεία καταστράφηκαν και 2 εκατομμύρια σπίτια καταστράφηκαν περίπου. Οπότε ε, και μόνο πάνω σε ανθρωπιστική βάση να το δούμε, ε, είναι συντριπτικά τα επιχειρήματα που συνηγορούν υπέρ της προσέγγισης αυτής. Είναι πραγματικά αυτή η ε, χαλάρωση των δεσμολογικών εμποδίων αναγκαία. Δεύτερον, μια πρόταση θα πω. σε σύγκριση με την ε, παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, το παρόν επίπεδο, δηλαδή η αύξηση των εισαγωγών, δεν θα υπερβεί το μισό τα εκατό και λιγότερο από μισό τα εκατό θα είναι η διαφορά λόγω της προτίμησης, της προτίμησης που θα δώσουμε. Δεν πρόκειται δηλαδή η χαλάρωση των ε, δασμών ε, να μας επηρεάσει εμάς. Ενώ για το Πακιστάν η διαφορά είναι πολύ σημαντική, θα βοηθήσει. Και μετά από αυτό θα ήθελα να ακούσω τους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Έχουμε οκτώ άτομα που ζητούν το λόγο. Πρέπει λοιπόν να σας ζητήσω να περιοριστείτε στα δύο λεπτά. Ευχαριστώ. 11 και κλείνω ο κατάλογος των ομιλητών. Τζαν Λούκα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ πιστεύω ορισμένα από τα θέματα που θέλω να θίξω εγώ, τα είπα ο συνάδελφος, θα τις υπάρχει ένα θέμα επί της ουσίας της χρήσης του εμπορίου για να έχουμε μια ανθρωπιστική παρέμβαση και για να υποστηρίξουμε ουσιαστικά τη συνεργασία με μια χώρα που βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση και με μια οικονομική και κοινωνική κατάσταση πραγματικά δυσχερή. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να κατανοήσουμε, να καταλάβουμε αν πρόκειται για μια κατεξαίρεση συμφωνία, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να είναι μια εξαιρετική συμφωνία αν εννοούμε τελικά προτιμησιακή γιατί σε όλες τις μεγάλες ε, περιοχές του κόσμου μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδεί θέματα διεθνούς πολιτικής, παγκόσμιες προκλήσεις, ε, Μπορούμε να έχουμε παραδείγματο χάρη το θρησκευτικό φονταμεταλλισμό ισλαμικού, ισλαμικής προέλευσης. Άλλη φορά, άλλες φορές έχουμε άλλες μορφές φονταμεταλλισμού ή ρατσισμού ή υπεριαλισμού ή νεοπικιοκρατίας. Έτσι λοιπόν κάθε φορά εμείς θα έπρεπε να διαφοροποιούμε ανάλογα με τις 27 ε, διαφορετικές πολιτικές ε, εξωτερικής άμυνας και ασφαλείας που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν εμείς αυτό πρέπει να το αποκαλέσουμε με το όνομά του. Είναι μια οικονομική παρέμβαση που ε, ουσιαστικά ευνοεί μια περιφέρεια στον κόσμο και φυσικά υπάρχει και το θέμα της ε, διεθνούς πολιτικής ασφάλειας, αλλά θα έπρεπε να ε, ε, οδηγήσει την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής να ασχοληθεί με αυτό και πρέπει ε, όλοι εμείς πρέπει να θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα θέμα που αφορά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 550 εκατομμύρια των Ευρωπαίων πολιτών και τα 27 κράτη-μέλη. Και όχι μόνο έναν οικονομικό τομέα, δηλαδή της φαντουργίας, όπου εμπίπτει το βάρος αυτής της επιλογής ε, αυτής τη διεθνού πολιτικής βοήθεια, γιατί αυτό είναι και αυτό είναι απαράδεκτο πέρα από οποιαδήποτε διαμεσολάβηση βρούμε και πιθανότατα θα το βρούμε ε, διασφάλιση, ρήτα διασφάλισης, αντιστάθμισης κτλ. Αλλά εμεί πρέπει να αναρωτιόμαστε και τελειώνω αν είναι δίκαιο ένα τομέα που από ε, 2,5 εκατομμύρια άτομα πρέπει να υποστηρίζει μια τέτοια πολιτική και δεν πρέπει να μιλάμε για πλέον ανθρωπιστική βοήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο από το ΕΛΚ. Συγγνώμη, Πρόεδρε. Εγώ συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με όσα το τον συνάδελφο Σούστα. Όλοι λυπούμαστε πολύ για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Πακιστάν και ο πληθυσμός του. Όμως εγώ νομίζω ε, αυτό μας οδηγεί στο να δώσει την απαραίτητη χρηματοοικονομική και ανθρωπιστική βοήθεια η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει το Πακιστάν αυτή η κατάσταση. Σίγουρα έχει δεσμευτεί απέναντι στον πακιστανικό λαό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει πάρα πολλέ οδού και μέσα για να ε, καταστήσει ε, αποτελεσματική αυτή τη βοήθεια. Τώρα, ε, αυτό που συζητούμε υπό τη μορφή επέκτασης καταβολής δασμών για τα επόμενα τρία έτη από την 1η του 2011 όμως θεωρούμε ότι δεν είναι ο πιο αποτελεσματικός μηχανισμός. Οι εμπορικές κορίσεις θα ωφελήσουν μόνο τους εισαγωγείς και τους εξαγωγείς και ε, εν τέλει επιχειρήσεις που στον τομέα της υφαντουργίας είναι εντατικού κεφαλαίου και ιδιαίτερα ανταγωνιστικές. Δεν θα ε, βοηθήσουν ε, τα άτομα ε, και τους τομείς που έχουν θυγεί άμεσα από τις πλημμύρες. Αυτοί χρειάζονται πολύ συγκεκριμένη βοήθεια και δύσκολο, δύσκολα θα τη λάβουν από αυτές τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Έτσι λοιπόν δεν κατανοούμε τι αντίκτυπο θα έχει ε, στον ε, Ευρωπα... Εμείς θεωρούμε ότι θα έχει μεγάλο αντίκτυπο ε, αυτό στην ευρωπαϊκή υφαντουργία, δηλαδή και στον ισπανικό τομέα αλλά και ε, στον τομέα της υφαντουργίας το 85% μιλάμε για τελειοποιημένα προϊόντα και για προϊόντα υφαντουργίας και εκεί τα ε, οι δασμοί των δεσμών φτάνουν το 12%. Έτσι λοιπόν, αν προβείτε σε αυτή ε, την ενέργεια, θα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη επίπτωση. Μάλιστα, άλλες χώρες όπως η Ιαπωνία δεν έχουν επιλέξει ε, τέτοια βοήθεια προς το Πακιστάν και αυτό θα μας θέσει σε μειονεκτική θέση. Επίσης, η Ινδία και το Μπαγκλαντές υποστηρίζουν τις εμπορικές παραχωρήσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριο Παύλο Σάλμπα. Κρίστοφερ Φιέλνερ, πάλι από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως θα ξέρετε συζητήσαμε και εσείς ε, και εγώ σε πολλές συζητήσεις στο θέμα. Είμαι υπέρ αυτής της πρότασης ε, και είμαι πολύ χαρούμενος που μπορούμε να συνδυάσουμε τη βοήθεια και το εμπόριο ούτω ώστε να μην δίνουμε με το ένα χέρι και αφαιρούμε αυτά που δώσαμε με το άλλο. Τώρα αν θυμάμαι καλά είναι κάτι το έκτακτο αυτό, το εξαιρετικό κατά έναν τρόπο, αλλά δεν είναι και εντελώ καινούριο, γιατί αν θυμάμαι καλά είχε γίνει κάτι τέτοιο προηγουμένως ε, με μονομερή διακοπή της ε, των και ε, για την ώρα έχουμε λάβει αυτό το μέτρο για να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη. Η αρχή την οποία υπογράψαμε ισχύει και για άλλους τομείς, γι' αυτό είναι σημαντικό να τη χρησιμοποιήσουμε και σε αυτόν τον τομέα. Από ό,τι καταλαβαίνω θα υπάρξει μια διαδικασία σύμφωνα με τη συνθήκη και αυτό θα το πούν και οι συνάδελφοι στο Στρασβούργο. Από ό,τι κατανοώ ορισμένες βιομηχανίες και ορισμένες χώρες ε, λένε ότι θέλουν να... Ε, το πληρώσουν αυτό, αυτή τη διαδικασία. Όταν το εξετάζω από τη δική μου προοπτική, κατά κάποιο τρόπο δεν μου φαίνεται παράδοξο το ότι ορισμένες βιομηχανίες θέλουν να πληρώσουν γιατί κατά κάποιον τρόπο ε, καλύπτονται από άλλους. Ε, αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Ε, ο Ντάνιελ εδώ μιλάει για μου κάνει νόημα ότι ξέρει μια τέτοια βιομηχανία. Εν πάση περιπτώσει είμαστε πολύ μακριά από το στόχο μας, ειδικά στον υφαντουργικό τομέα. Και ε, νομίζω ότι πρέπει να μπορούμε να δίνουμε, πρέπει να δίνουμε μάλλον όταν μπορούμε. Και είχαμε αποφασίσει να δώσουμε όσο περισσότερα γινόταν ε, για τον αγωγό φυσικού αερίου παραδείγματος χάρη. Λοιπόν, ελπίζω ότι θα είμαστε σύντομοι, ότι αυτή η διαδικασία θα είναι γρήγορη. Δηλαδή δεν θα πρέπει να ξαναλέμε τα ίδια δύο χρόνια μετά. Αν κάνουμε κάτι να το κάνουμε τώρα και γρήγορα. Αυτό είναι και το κυριότερο σημείο από όλα πιστεύω. Ο Μάριο από το ΕΛΚ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επανέλθω στα επιχειρήματα τα οποία υπέβαλαν οι άλλοι συνάδελφοι που μίλησαν κατά των προτάσεων της Επιτροπής, συναξάπαντες. Ε, τώρα επιμένω με ε, περιμένω με ανυπομονησία την απάντηση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή να δούμε τι μέτρα θα ληφθούν, τα κατεπήγοντα αυτά μέτρα που θα προβλέπονται για τρία χρόνια. Πρώτον, αν μπορούσα να προσθέσω ένα στοιχείο το οποίο δεν αναφέρθηκε μέχρι στιγμής, δεν κατανοώ γιατί, καθόλου δεν κατανοώ, ότι υπάρχει για τη ζάχαρη ε, ποσοστοποίηση, γιατί για τα άλλα προϊόντα δεν μετρούμε καθόλου τις ποσότητες, οπότε... Ε, ίσως για προϊόντα της ίδιας προέλευσης με τη ζάχαρη να μπορεί να γίνονται μόνο καταμετρήσεις. Λοιπόν δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Μπορεί να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιε θα είναι οι επιπτώσεις. Δεν ψηφίζουμε μέχρι να τις έχουμε. Χωρίς επιπτώσεις πώς θα ε, λάβουμε αποφάσεις. Ε, ο εισηγητής ο οποίος προέρχεται με μια, από μια χώρα η οποία έχει δυσκολία με αυτά τα μέτρα, μέτρα που αφορούν τις εισαγωγές, νομίζω ότι θα πρέπει να ενθουσιαστεί από αυτήν την πρόταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Στέντι. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι θα πιστεύατε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει μόνο όφελος από αυτή τη διαδικασία γιατί εγώ ήμουνα στην ε, βιομηχανία την, της υφαντουργίας, Έχει, είχε μεγάλη βιομη, μεγάλες βιομηχανίες υφαντουργίας, τώρα όλα αυτά εξαφανίστηκαν και τώρα είμαστε σχεδόν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε μικρή επίπτωση ό,τι και να κάνουμε ούτως ή άλλως. Συμφωνώ απόλυτα με τον Κρίστοφερ, με όλα όσα είπε. Ε, νομίζω ότι όλη την ημέρα, σήμερα, το μεγαλύτερο κομμάτι της μέρας μιλούσαμε για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τη χρηματοοικονομική κατάσταση και ένα από τα όπλα μας είναι το εμπόριο με άλλες χώρες. Όταν μιλάμε για το φυσικό αέριο έχει καταστροφικά αποτελέσματα τόσο πολύ που θέλουμε να σταματήσουμε το εμπόριο. Ε, με την αντίστοιχη χώρα. Που θα ήθελα να εξετάσουμε από κοντά, πάντα το πίστευα αυτό, το εμπόριο, το ίδιο το εμπόριο και όχι τις βοήθειες και τη στήριξη. Και νομίζω και ότι ο εισηγητής πιστεύει τα ίδια με μένα. Ο, ε, η, η Χωσέ Ανδρέας, ναι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η αλήθεια είναι ότι είναι απαραίτητες αυτές οι ενισχύσεις ε, στις χώρες ε, που υποφέρουν και εγώ νομίζω ότι τέτοια βοήθεια συμπεριλαμβάνεται σε πάρα πολλές διεθνείς συμφωνίες, δηλαδή κατάργηση των δεσμών ε, προκειμένου να βοηθήσουμε την υφαντουργία και την παραγωγή μιας χώρας στον τομέα αυτό όμως σε αυτές τις συμφωνίες και συγκεκριμένα συμφωνία με το Πακιστάν έχει αρνητικές συνέπειες για συγκεκριμένους τομείς όπως συγκεκριμένα είναι η φαντουργία για την οποία συζητήσαμε εδώ, το είπαν και άλλοι συνάδελφοι. Αυτά οι επιπτώσεις θίγουν κυρίως χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία και θα πω ένα αριθμητικό στοιχείο. 16% των ε, συναλλαγών της Ισπανίας προέρχεται από την φαντουργία και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό νούμερο όπως βλέπετε. Εγώ πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Αγορά Υφαντουργίας έχει κάποιες ε, ζώνες ε, που μπορούμε εμείς να πουλήσουμε στη Γαλλία και στη Γερμανία δηλαδή. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να αποφύγουμε να ε, έχουμε αρνητικές συνέπειες στην απασχόληση αλλά και στην παραγωγή και έχουμε και την πρόταση του Βελγίου να μειώσουμε την περίοδο 2-3 ετών για να δημιουργήσουμε μηχανισμούς εποπτείας και την δυνατότητα να έχουμε ποσοστώσεις το δεύτερο έτος από το 2012 βάσει μελέτης που θα γίνει γίνει το 2011. Εγώ νομίζω ότι είναι λογική αυτή η πρόταση, εφόσον θα έχουμε μία αξιολόγηση κάθε τέσσερι μήνε και θα αξιολογούμε τον αντίκτυπο. Νομίζω ότι θα ήταν λοιπόν κάτι θετικό, αλλά πάντοτε διασφαλίζοντα και προστατεύοντα και τι δικέ μα θέσει εργασία και τη δική μα βιομηχανία. Ευχαριστώ, Ωσέφα. Τώρα ο κ. Μαργκάντη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ είμαι υπέρ ε, στο να βοηθήσουμε το Πακιστάν, αλλά είμαι εντελώς αντίθετο στην πρόταση αυτή. Εδώ ε, γνωρίζουμε ότι ε, πλήγησαν ε, και περιοχές που βρίσκονται και πιο απομακρυσμένα από το ποτάμι. Μεγαλύτερες ζημιές έγιναν επί των καλλιεργειών και επί της αγροτικής παραγωγής. στο Πακιστάν πολλές φορές προσέφυγε στις ενισχύσεις και στην κατάργηση των δασμών, αλλά πάντοτε Αυτό ε, έγινε με πάρα πολλές ε, ε, αιτίε, δηλαδή έγινε και για την καταπολέμηση τρομοκρατίας και τώρα το ζητά για τις πλημμύρες. Το Πακιστάν ήδη καλύπτεται από ένα σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων και το 60% σχεδόν των εξαγωγών του προς την Ευρωπαϊκή Ένωση την χάνει χαμηλότερων δασμών και ένα μεγάλο ποσοστό και μηδανικών δασμών. Έχουν ήδη δοθεί ενισχύσει στο Πακιστάν. Εγώ με της είμαι μέλο τη επιτροπή Προπολογισμού, με συγχωρείτε, και μεταφέραμε μάλιστα και 50 εκατομμύρια φέτος, ενώ άλλες χώρες ε, θα πληρώσουν πάλι στο Πακιστάν ένα ε, πολύ μεγάλο ποσό ενισχύσεις και από το 2005 συγγνώμη, μιλήσαμε για το 0,5% ε, ε, επίπτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως αυτή η επίπτωση θα είναι σε τρία κράτη-μέλη, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία. Και εγώ θέλω να ήξερα ποιος θα αποζημιώσει αυτά τα κράτη. Είναι λοιπόν ε, σωστό να δώσουμε τη βοήθεια, αλλά όλα τα κράτη ισότιμα να συμμετέχουν σε αυτή την βοήθεια, στην έργη βοήθεια. Ε, ε, τι μπορώ να σα πω ότι εγώ ειλικρινά είμαι αντίθετο με τον τρόπο χορήγηση αυτή τη βοήθεια. Αρήφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ειλικρινά, πέρα από το αποτέλεσμα που θα προκύψει, σε σχέση με το αν θα συμφωνήσουμε ή όχι από της πρότασης, να σας πω ότι με εκπλήσει η πρόταση που γίνεται από το Συμβούλιο και που θα τη εφαρμογεί η Κομισιόν. Γιατί, γιατί δεν μπορούσαμε να ανταποκριθούμε, να απαντήσουμε σε μία ε, ανθρωπιστική ε, κρίση. Και εδώ, ε, τι να σας πω, φαίνεται ότι προσπαθούμε να βρούμε ένα, ένα τρόπο να απαντήσουμε για το Πακιστάν έκτακτα. Τώρα, εδώ μας δίνεται και μία εικόνα αλλοιωμένη σε σχέση με το την Ευρωπαϊκή Ένωση και ανάλογα ε, με το ποια είναι η χώρα η οποία θίγεται, φαίνεται να μπαίνουμε εμείς σε συγκρούσεις. Ε, ακούσαμε και τον Βρετανό φίλο, ο οποίος... Ε, ε, είπε ότι φαίνεται ότι υπερασπίζεται τους Πακιστανούς υπηκόους. Εγώ νομίζω ότι με τέτοιες προτάσεις δίνουμε πάρα πολύ κακή εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να είμαι ειλικρινής. Τρίτον, πρέπει να μας πείτε αν ε, ε, πρόκειται για μια βούληση η οποία έμεσα μεταφράστηκε κατά αυτόν τον τρόπο για να έχουμε κάτι παραπάνω που δεν μπορούμε να το αποκτήσουμε μέλα μέσα ή να μας εξηγήσετε ποιες είναι οι επιπτώσεις για την στρατηγική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διεθνές επίπεδο και το εμπόριο θα είναι αυτό. Αλλά κανείς δεν μας παρουσίασε αυτά τα στοιχεία. Έτσι λοιπόν... Εγώ να σας πω ότι είμαι πολύ σόφρον, αλλά ε, είμαι και πάρα πολύ ευαίσθητος και θέλω να ε, βοηθούμε σε περιπτώσεις ανθρωπιστικής κρίσης ε, και εγώ θα ήθελα να μην τίθεται εδώ θέματα ότι ο τάδε συνάλφος λέει ε, αυτά τα πράγματα επειδή προέρχεται από την ε, Δίνα χώρα. Μήπως δεν θα υπήρχε κάποια άλλη λύση ε, ε, μήπως ε, να απαντήσουμε στην ε, ανάγκη του Πακιστάν με άλλο τρόπο. Δηλαδή γιατί να μην δώσουμε μία μακροοικονομική βοήθεια. Στο παρελθόν έχει γίνει κάτι γιατί να μην βρούμε παραδείγματος χάρη γραμμές προπολογισμού για την ανθρωπιστική βοήθεια κτλ. Εγώ νομίζω ότι εδώ λοιπόν συλλογικά πρέπει να αγγιόμαστε για την εικόνα που δίνουμε στο εξωτερικό για να μην φαίνεται ότι έρχονται ερχόμαστε εδώ να υπερασπίσουμε ε, τα εθνικά μας συμφέροντα και δεν είμαστε γενναιοδοροί απέναντι στο Πακιστάν. Ευχαριστώ. Κύριε Τσέλεφ, από τους Πρασίνους. Uh, uh. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μιλώ εξ ονόματος των Πρασίνων. Είμαι σκιώδης για το θέμα. Οι πράσινοι υποστηρίζουν τη χαλάρωση των ε, δασμών, των προτιμήσεων αυτών για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Δεν θα θεωρηθεί αυτό πύλη που θα αλλάξει το καθεστώς ε, GSP-SYN. Το Πακιστάν έχει πολύ δρόμο να κάνει μέχρι να πληρώσει τις ε, απαιτήσεις του συστήματος Τώρα, για να δούμε καλύτερα τα 75 προϊόντα που αναγράφονται. Εγώ άκουσα τους παραγωγούς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Πακιστάν και καταλαβαίνω κάποιες ανησυχίες που εκφράστηκαν. Θα προέτεινα να σκεφτούμε τη συνολική αξία των πρόσθετων προϊόντων που θα έρχονται στην Ευρώπη και που, θα, που εκτιμώνται σε 100 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Σκέφτομαι μήπως θα μπορούσαμε να βάλουμε μια αξία σε κάθε σειρά προϊόντος, γιατί αυτό θα ε, καθησύχαζε κάποιους φόβους από, που έχουν οι παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ίσως υπάρχει και κάποια παρεξήγηση γιατί η άδεια για την εθανόλη για εισαγωγή 100.000 τόνους το χρόνο ε, έχει σχέση, συσχετίζεται με το αβιοκαύσιμα, αλλά δεν είναι μετουσιωμένη, ε? ειναι undenatured, είναι μη μετουσιωμένη εθιλική αλκοόλη. Άρα θεωρώ ότι είναι για ανθρώπινη κατανάλωση. Δεν θα χρησιμοποιηθεί αυτή ως βιοκαύσιμο. Επιβεβαιώστε μου παρακαλώ, γιατί βέβαια οι πράσινοι δεν θα ήθελαν αύξηση των βιοκαυσίμων που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να διαβεβαιωθούμε ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο και ότι η μη μετουσιωμένη εθιλική αλκοόλη θα πάει για ανθρώπινη κατανάλωση. Σύντομα παρακαλώ, συντομεύεται. Αυτά είχα να σας πω. Τελείωσα κιόλας. Από την ομάδα του ΚΟΕ, Χάρολτ Σούλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύμφωνο με πολλές επικρίσεις που εξέφρασαν οι συνάδελφοι στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων για τη διαδικασία rollover από το GSP-SYN ε, είχαμε συμφωνήσει για κάποια προβληματική που έθιξα και εγώ και υπήρχε ε, ενιαία απόψη όλων των πολιτικών ομάδων ότι αυτό δεν θα έπρεπε καν να το εξετάσουμε, δηλαδή η σύνδεση της ανθρωπιστικής βοήθειας, της βοήθειας έκτακτης ανάγκης με τη διαδικασία ε, GSP SIM και τώρα πάλι βλέπουμε αυτό το σημείωμα της Κομισιόν που μας κάνει να αναρωτιόμαστε τι είναι αυτό τώρα, αυτή η νέα έμφαση που δίδεται εδώ. Ο συνάδελφος Σούστα έχει δίκιο νομίζω ότι πρέπει καταρχήν να δούμε ποιοι είναι οι κλάδοι που θίγονται άμεσα, ποιες πληθυσμιακές ομάδες ε, δεν θα αντιμετωπίσουν δεν θα μπορέσουν να κάνουν πάλι οικονομική δραστηριότητα μετά τις πλημμύρες. Ε, ακούσαμε ότι η πακιστανική κυβέρνηση, οι πακιστανικές αρχές και οι περιφερειακές δομές χρειάζονται ανασυγκρότηση και ε, ανοικοδόμηση 2 εκατομμυρίων κατοικιών ώστε να είναι ανθρώπινες οι συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού. Και ερωτώ την Κομισιόν, Ποιες συγκεκριμένες προτάσεις υπάρχουν ούτως ώστε να ανταποκριθούμε σε αυτό το θέμα και να φροντίσουμε για την επιτόπια παραγωγή με κάποια και κάποια οικονομική και εμπορική δραστηριότητα. Πώς θα τους ε, ε, υποστηρίξουμε. Τώρα για την εθανόλη. Δεν είναι μόνο ε, οι ανησυχίες των πρασίνων εδώ που είναι σημαντικές, αλλά γενικότερα τίθεται το θέμα μετά τις πλημμύρες δεν θα έπρεπε να προβλεφθούν καλλιέργειες τροφίμων, ε, καλλιεργιών που θα ε, καταναλωθούν ως τρόφιμα. Ε, επίσης να ρωτήσουμε συγκεκριμένα τις πακιστανικές αρχές ποιες κλάδ, ποιους κλάδους θα ενισχύσουν στην πακιστανική οικονομία. Αυτές ήταν οι παρατηρήσεις μου και ευχαριστώ. Ο κύριος Κάσπαρη από το ΕΛΚ. Αγαπητοί μου συνάδελφοι, Σήμερα μιλήσαμε μόνο για τις χώρες παραγωγούς που θίγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα διατεθούν χρήματα θα διατεθούν χρήματα και από τους 27 και από τους net payers. Ε, κάποιοι ε, θα επηρεαστούν μέσω της κλωστοϊφαντουργίας, άλλοι μέσω της ε, καθαράς συνεισφοράς τους. Πάντως η Κομισιόν δεν παρουσίασε επαρκώς τις θετικές επιπτώσεις για το Πακιστάν. Οι εξαγωγές λέτε ότι από 900 θα εκατομμύρια θα πάνε σε ένα δις. Μια αύξηση εξαγωγών κατά 100 εκατομμύρια ευρώ δηλαδή. Από την άλλη πλευρά χάνομαι... Ε, 80 εκατομμύρια ευρώ από τις ε, ειδικές αυτές, ε, τα ειδικά έσοδα. Μήπως θα ήταν καλύτερο, αντί για ένα, δύο, τρία χρόνια να μειώσουμε τις δασμολογικές γραμμές, ε, μήπως πιο καλό θα ήταν τα 80 εκατομμύρια έσοδα να μην τα πάρουμε και να τα δώσουμε στο Πακιστάν. Καλό θα ήταν να μας πει η Κομισιόν πώς το βλέπει αυτό. Επίσης, γιατί λέει Άστον και όλη η διοίκηση δεν ασχολήθηκε με το θέμα, γιατί αυτά είναι εξωτερική πολιτική. Περισσότερο είναι θέματα στρατηγικής, όχι τόσο εμπορικά. Καλό θα ήταν η Βαρόνη Άστον, να πάρει σαφή θέση και να πει ότι ε, αφού η Κομισιόν δεν θεωρεί τόσο σημαντικό το θέμα, παίρνουμε αμέσω θέση εμείς. Νομίζω πάντως ότι θα έπρεπε να πιστούν οι συνάδελφοι και η Κομισιόν. Καλό είναι να μας πει τι ακριβώς θέλει και να μας το παρουσιάσει αυτό σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο. Ε, ας ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Έχουμε πέντε λεπτά. Ποιος θέλει να λάβει το λόγο. On of this Για αυτήν την ε, πρωτοβουλία και για το που, ε, προς τα που κατευθύνεται. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέγομαι Πίτερ Μπέτς ε, και δουλεύω στην Γενική Διεύθυνση 3 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την ανταλλαγή απόψεων, για αυτή την πολύ επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων και χαίρομαι που θα δουλέψω μαζί με τον εισηγητή. Πραγματικά είναι μια καταστροφή τεράστια στο Πακιστάν. Δεν ε, ε, περατώθηκε μεν η καταστροφή αλλά οι επιπτώσεις θα είναι παρούσες για πάρα πολύ καιρό δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω τα πράγματα υπάρχουν απώλειες χωρίς προηγούμενο και βεβαίως χρειάζονται και μέτρα χωρίς προηγούμενο το ε, εμπόριο επίσης πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσουμε μια τέτοια φρικτή κατάσταση σε μια χώρα που ε, υποφέρει. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έκανε μια διακήρυξη στις 16 Σεπτεμβρίου. Ε, αναγνώρισε ότι το εμπόριο θα πρέπει να είναι μέρος ενός πακέτου μέτρων βραχυπροθέσμων, μεσοπροθέσμων και μακροπροθέσμων μετά στα οποία είναι και η ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό είναι ένα πακέτο το οποίο ε, συμπεριλαμβάνει το εμπόριο. Αυτό αναγνωρίστηκε με μεγάλη σαφήνεια. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αυτά τα μέτρα που είναι πάρα πολύ φιλόδοξα για την οικονομική ανάκαμψη και την αύξηση θα πρέπει να φορούν ειδικά το Πακιστάν και να πάρουν το, τη μορφή των, της μείωσης των φόρων Πρέπει να είναι άμεσα, θα πρέπει να είναι συμβατά με άλλες αποφάσεις που θα λαμβάνουν ε, υπόψη τις ανάγκες της ε, στιγμής. Είναι σχεδόν αδύνατη η επιτέλεση αυτού του έργου γιατί έχουμε μία πρόταση καλέσαμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να παρουσιάσει κάποια πρόταση ήδη από τον Οκτώβριο και μέσα σε τρεις εβδομάδες πρέπει να παρουσιάσουμε αυτήν την πρόταση η οποία προσπαθεί να τετραγωνίσει τον κύκλο με τις παραμέτρους που διαθέτουμε. Η πρόταση αυτή είναι ε, μία πρόταση για 75 προϊόντα, γραμμές προϊόντων. Πώς θα μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε και τα 75. Πρέπει να δούμε τις παραμέτρους του Ευρωπαϊκού ε, ε, Συμβουλίου για το ε, input κλειδί πρέπει να πούμε ότι είναι κάπως εύκολο στη συνέχεια να προχωρήσουμε, να το αφαιρέσουμε από την, τον κατάλογο των ε, προϊόντων για τα οποία δεν πληρώνει δασμού στην εισαγωγή το Πακιστάν. Στη συνέχεια θα πρέπει να αφαιρέσουμε όλα εκείνα τα προϊόντα που υπάγονται στις ε, προτιμήσεις σύμφωνα με τη Γενική μου Διεύθυνση. Υπάρχουν επίσης ε, ε δασμοί anti-dumping για ορισμένα chips που είναι πάρα πολύ φτηνά ε, υπάρχουν επίσης και άλλα προϊόντα που απομένουν που διευκολύνουν την εξαγωγή ε, ορισμένων σκευών, παραδείγματος χάρη, που τα χρησιμοποιούσε το Πακιστάν για, να, για τροφή, για να τρέφει ανθρώπους. Ε, και ε, χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε συνολικά τη βιομηχανία με κάποια ευαισθησία. Υπάρχουν ορισμένες μεγάλες μάρκες όπως η μάρκα B που είναι, ε, κάνει τεράστιες εισαγωγές. Έχουμε ένα αποτέλεσμα 25 προϊόντων όλων των 25 γραμμών για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, τι είναι δυνατό να γίνει. Ε, υπάρχει ας πούμε στον υφαντουργικό τομέα το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης και όλες οι, ένα 25% των εξαγωγών του Πακιστάν υπάγονται σε αυτόν τον τομέα. Όλες λοιπόν οι εξαγωγές ε, χωρίζονται σε διάφορα προϊόντα, μερικά από τα οποία είναι προϊόντα κλειδιά. Υπάρχουν ορισμένα τέσσερα προϊόντα, έξι ε, που έχουν σχέση με το δέρμα ε, και τροφή, ορισμένα μανιτάρια για παράδειγμα, ε, φιλελευθερωποίηση 74 προϊόντων προτείνεται και ποσοστώσεις για ε, ορισμένα άλλα. Αυτό θα είναι το τελικό αποτέλεσμα που θα αφορά το 27% των εισαγωγών των ε, τρεχουσών εισαγωγών του Πακιστάν και μέσα στις προοπτικές είναι τα Έχουμε 100 ε, εκατομμύρια το χρόνο τα οποία αναμένουμε να εισπράξουμε. Ε, για τις 75 γραμμές προϊόντων είναι 18 δισεκατομμύρια. Ε, στα 15 ε, δισεκατομμύρια προσθέτουμε και άλλα 100 εκατομμύρια. Οπότε τελικά έχουμε μία μείωση των εισαγωγών και μία μείωση της παραγωγής αυτά τα 75 ε, προϊόντα και τα 100 εκατομμύρια για τα οποία σας μίλησα. Τρία χρόνια είναι η διάρκεια, εμείς προτείναμε δύο χρόνια για να είμαστε αξιόπιστοι, γιατί έτσι ήταν η αρχική μας πρόταση και τελικά πρέπει να πάμε στην Γενέβη και πρέπει αυτό να γίνει μόνο για το Πακιστάν όπως προσδιορίζει η εντολή μας και μπορείτε να φανταστείτε τι συζητήσεις θα έχουμε στη Γενέβη, πόσο δύσκολες θα είναι και τι επιπτώσεις θα έχουν για τους ανταγωνιστές του Πακιστάν. Έχουμε αναλάβει τη δέσμευση, εν πάση περιπτώσει, να θεσπίσουμε ορισμένα κριτήρια Βεβαίω δεν ξέρουμε πόσο πρακτικά είναι αυτά τα κριτήρια και σε τι ανταποκρίνονται ακριβώς και νομίζω ότι πληροφόρησε σωστά την Επιτροπή για τη δυσχέρεια της κατάστασης. Ευχαριστώ πολύ. Πέρα στη συζήτηση. Ε, είδατε ότι η Επιτροπή δεν μπόρεσε να απαντήσει σε καμία από τις ερωτήσεις που θέσαμε σε σχέση με αυτό το θέμα. Το παρατηρήσατε αυτό. Θα να βάλουμε το 19 και το 20 ούτω ώστε να μπορέσουμε να περατώσουμε την ημέρα μας και να φύγουμε ήσυχοι. Ένα μεγάλο μέρος είναι, έχει τελειώσει τη συνεδρίασή μας. Παρακαλώ να φύγουν όλοι από την αίθουσα εκτός από τους συντονιστές. Μόνο αυτοί που θα πάρουν μέρος στη συνάντηση των συντονιστών θα παραμείνουν. Όλοι οι άλλοι, παρακαλώ, εξέλθετε χωρίς πολλές συζητήσεις και θόρυβο.